Συγγνώμη για την τρίλεπτη καθυστέρηση, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα προσπαθήσω να βελτιωθώ στο μέρο. Εδώ ήμουν, αλλά άκουγα κάποιου Ιρλανδού που μιλούσαν για την οδική ασφάλεια. Επόμενο είμαι στην ημερήσια διάταξη. Έκθεση Τσικάου για υπογραφή και σύναψη συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδά για την ασφάλεια τη πολιτική αεροπορία. Σίλβια, έχει και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μιλούμε για την απόφαση Συμβουλίου και Επιτροπή ότι αφορά τη σύναψη συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωση και Καναδά για την ασφάλεια τη πολιτική αεροπορία. Υπάρχει και μια συμφωνία πλαίσιο για τις αερομεταφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά. Η τελευταία συμφωνία αφορά την ασφάλεια στην πολιτική αεροπορία. Οπότε έχουμε δύο διαφορετικές συμφωνίες. Η συμφωνία πλαίσιο πρέπει να επικυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη. Πάντως, η συμφωνία αυτή για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας θα πρέπει να εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά δεν χρειάζεται να κυρωθεί και από τις 27 χώρες μέλη. Μέχρι στιγμής μόνο 6 χώρες μέλη έχουν διμερείς συμφωνίες με τον Καναδά για την πιστοποίηση προϊόντων και η νέα συμφωνία θα αντικαταστήσει αυτές τις 6 διμερείς συμφωνίες. Η νέα αυτή συμφωνία θα ισχύσει και στις 27 χώρες μέλη και έχει χονδρικά την ίδια δομή με τις υπάρχουσες συμφωνίες για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Πρόκειται για υποδειγματική συμφωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς έχουν πολύ πυκνές αερομεταφορές και κατασκευάζουν και αεροσκάφη. Γι' αυτό και οι διαδικασίες πιστοποίησης είναι πολύ σημαντικές. Με την τελευταία συμφωνία απλουστεύεται η κατάσταση και περιορίζεται η γραφειοκρατία. Μάλιστα, η επικάλυψη ελέγχων και αξιολογήσεων θα περιοριστεί στο ελάχιστο και οι δύο, τα δύο συμβαλόμενα μέρη, Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδά, θα στηρίζονται στα αμοιβαία τους συστήματα πιστοποίησης. Μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ των συμβαλωμένων μερών θα ελεγχθεί κατά πόσο τα εμπλεκόμενα σώματα είναι ικανά να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Και μάλιστα θα συσταθεί και μια επιτροπή για να προτείνει λύσεις για ενδεχόμενα προβλήματα. Και παραλαμβάνω ότι η συμφωνία είναι περίπλοκη, υποδειγματική, πολύ ισχυρότερη πολύ καλύτερη από... και πληρέστερη από άλλες συμφωνίες που έχουν συναυθεί διμερώς με χώρες. Εμείς θα προτείνουμε την έγκριση αυτής της ε, συναψυμφωνίας. Με την συνθήκη της Λισαβόνας άλλαξε η νομική βάση και έγιναν οι απαραίτητες αλλαγές και στη διαδικασία. Η διαδικασία ξεκίνησε μετά τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας και όλες ε, οι αλλαγές που έγιναν με τη συνθήκη ελήφθησαν υπόψη για τη σύναψη της συμφωνίας που μπορεί πλέον να αριστικοποιηθεί. Αυτά κύριε Πρόεδρε και περιμένω τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστούμε κυρία Τσικάου. Θα ήθελα να σας πενθυμίσω, συνάδελφοι, ότι με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνα απαιτείται συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά δεν προβλέπεται δικαίωμα τροποποίησης ε, του κειμένου της συμφωνίας. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αρνηθούμε τη συγκατάθεσή μας. Δηλαδή να δεχτούμε ή να απορρίψουμε τη συμφωνία, αλλά όχι να την τροποποιήσουμε. Αυτό έπρεπε να το είχα πει από την αρχή τη συζήτηση, αλλά τώρα το θυμήθηκα. Ο κύριο Κούν Από πλευράς Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο τι ευχαριστίε μας στην εισηγήτρια που επεξεργάστηκε το θέμα. Γνωρίζουμε ότι πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς την κατεύθυνση μια κοινή δράσεως της Ευρώπης απέναντι σε τρίτες χώρες. Έξι χώρες μέλη έχουν συνάψει ξεχωριστή συνθήκη σχετικά με ε, μια συμφωνία για την αεροναυσιπλοεία μαζί με τον Καναδά, είναι σωστό που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία Κομισιόν να επεκτείνει την συμφωνία αυτή σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, κάτι το οποίο θα έχει σχέση και με την πιστοποίηση των αεροσκαφών, αλλά και των δομών ασφαλείας. Συνεχίζονται εντατικά οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων των εμπορευμάτων και των επιβατών με τον Καναδά. Είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα με τις Ηνωμένε Πολιτείες γιατί έχουν πολύ αυστηρούς κανόνες σε ό,τι αφορά τη μεταφορά υγρών και φορτίου γενικότερα. Πάντως είναι καλό ότι έχουμε προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα. Θέλουμε και εμείς να δηλώσουμε ότι ως Λαϊκό Κόμμα θα εγκρίνουμε την ε, συνθήκη. Όπως είπε πριν ο πρόεδρος ε, Σίμψον, δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Δηλαδή είτε την δεχόμαστε είτε την απορρίπτουμε. Αλλά νομίζω ότι έχει γίνει σωστή δουλειά. Και σε ό,τι αφορά την Λισαβόνα, εμείς θεωρούμε καλό ορθό βήμα προς μια κοινή ευρωπαϊκή κατεύθυνση και θα πρέπει να ισχύσει σε όλες τις χώρες μέλη. Σας ευχαριστώ και πάλι για την προσπάθεια που καταβάλατε ως Μάισνερ. Ευχαριστώ. Πρόκειται για κάτι το νέο, το είπε και η κυρία Τσιγάου και την ευχαριστώ για την εργασία της. Είναι νέα η αρμοδιότητα αυτή για το Κοινοβούλιο. Δεν είναι τόσο εκτεταμένη όσο θα θέλαμε. Μπορούμε να πούμε μόνο ναι ή όχι, όπως είπε ήδη ο Πρόεδρος. Ωστόσο πρόκειται για σημαντική πρόοδο, ότι δηλαδή τώρα ακούγεται η φωνή μας. Και αυτό είναι το μέγα πλεονέκτημα που προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνος. Ότι δηλαδή τώρα ακούγεται τη φωνή του Κοινοβουλίου σε όλα τα νομοθετήματα και γνωμοδοτεί. Και βέβαια εμείς οι φιλελεύθεροι είμαστε υπέρ τη υπογραφής της συνθήκης αυτής διότι είναι σκόπιμη. Δεν είναι μονάχα έξι χώρε. δεν θα είναι μονάχα έξι χώρε, αλλά 27 χώρε οι οποίες θα κληθούν να εφαρμόσουν ε, την συμφωνία αυτή, που θα αντικαταστήσει τι επιμέρου ε, διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίε και ταυτόχρονα αποτελεί και μια κοινή τράπεζα διαπραγματεύσεων για την επίλυση προβλημάτων όπως αυτά που έθιξε η, η Και αυτό λοιπόν είναι σκόπιμο, εφόσον με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αποφύγουμε τις επικαλύψεις και η Ευρώπη ζει από τις εμπορικές συμφωνίες με άλλες χώρες. Ορθό λοιπόν που γίνεται αυτή η συμφωνία για την αεροναυσιπλοεία και ευχαριστούμε και πάλι την η ο κύριος Κράμερ των Πρασίνων. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ που είναι η συγγετριά μας είναι απούσα, αλλά ευχαριστούμε και εμείς για την εργασία της στην εισηγήτρια και θα υποστηρίξουμε. Με τον τρόπο αυτό θα αρθούν οι διμερείς συμφωνίες και θα αντικατασταθούν από αυτή τη συνολική ε, συμφωνία που όπως, είπα, όπως είπαν και άλλοι μάλλον είναι σκόπιμο. Είναι δύσκολο να βρεθούμε σε απόλυτα ισότιμη σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε, διότι οι Ηνωμένε Πολιτείε εκμεταλλεύονται ε, κάθε φορά τον κατακαιρματισμό της Ευρώπης και ένα αεροπλάνο που πηγαίνει από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορεί να συνεχίσει μεταφέροντας ε, φορτία ή επιβάτες μέχρι τον Άγιο Φραγκίσκο. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την εισηγήτρια, όπως και προλαλήσαντες για την συμφωνία αυτή με τον Καναδά. Εγώ είμαι και πρόεδρος της αντιπροσωπείας ε, για τη σχέση με τον Καναδά και με αυτήν την ιδιότητα χαίρομαι ιδιαίτερα για την συμφωνία. Βέβαια, στο μέλλον δεν ξέρω πώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εμπλέκει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαπραγματευτική διαδικασία, αλλά αυτό αφορά περισσότερο το μέλλον. Και μια και έχουμε πολλέ παρόμοιε συμφωνίε που θα κληθούμε να εξετάσουμε, καλύτερη συμμετοχή μας ε, να συζητηθεί έγκαιρα αυτή τη φορά, γιατί έχουμε νέες αρμοδιότητες με τη συνθήκη της Λισαβόνας και θα πρέπει να τις ασκήσουμε. Δεν θέλουμε να μας φέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτο τελεσμένο γεγονότος και να πρέπει μόνο να πούμε ναι ή όχι, αλλά να εμπλεκόμαστε σε νωρίτερο στάδιο της διαπραγματευτικής διαδικασίας και όχι μόνο στις ε, συμφωνίες πολιτικής αεροπορίας, αλλά σε όλες τις εμπορικές συμφωνίες με τις τρίτες χώρες. Πάντως, ό,τι αφορά την έκθεση Τσικάου και τη σύστασή της, ε, συμφωνώ απόλυτα ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του για την συμφωνία με τον Καναδά. Ωραία. Έχουμε τον κύριο Μπουργκέλη Βενέ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και να ευχαριστήσω βεβαίως και την κυρία Τικάου για την ε, έκθεσή της και τις συστάσεις, την σύσταση που απευθύνει προς την Επιτροπή σας, δηλαδή ότι το Κοινοβούλιο ε, να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του όσον αφορά την σύναψη αυτή τη ε, συμφωνία. Και να ευχαριστήσω και τα μέλη τη Επιτροπή σα που κατά την ίδια έννοια τοποθετήθηκαν ε, στα προλίγου. Όπω είπε και η κυρία Τικάου, είναι μια πάρα πολύ σημαντική ε, συμφωνία. Μπορεί να θεωρηθεί μάλιστα παραδειγματική σημασία, μια και καθορίζει πιο εύκολες εμπορικές ε, σχέσεις ανάμεσα ε, σε δύο μεγάλους κατασκευαστές ε, αεροπορικών συστημάτων, οχημάτων κλπ. Είναι σημαντικό να υπάρχει αμοιβαία αποδοχή και πιστοποίηση των διαδικασιών και εάν είναι δυνατόν ε, να υπάρχουν ε, ταυτόσημα πιστοποιητικά ε, πραγματικά αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κατασκευή των αεροσκαφών, των κινητήρων και των λοιπόν συστημάτων και πιστεύω ότι θα έχουμε κερδίσει και χρήμα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε μια μεγάλη ανταγωνιστική αγορά και ευχαριστώ την κυρία που το υπογράμμισε στην οι οικονομικές σχέσεις όσον αφορά τις ανταλλαγές αεροναυτικών προϊόντων και εξαρτημάτων μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης φτάνει στα 50 δις ε, ευρώ και επομένως ε, ε, είναι πάρα πολύ θετική η προσέγγιση αυτή ε, και είναι μια προσέγγιση η οποία, της οποίας κύριο μέλημα παραμένει η ασφάλεια. Ευχαριστούμε πολύ για τα όσα είπατε και για την θέση που πήρατε υπέρ της συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Τικάου, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που δέχτηκαν την θέση μας. Να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, πρότασή της αλλά και για τις πληροφορίες που έδωσα στη διάθεσή μας στην αρχή της εργασίες μας. Είναι βέβαιο ότι και οι καναδέζικες εταιρείε και οι ευρωπαϊκές θα κερδίσουν πολλά χρήματα μέσω της αμοιβαία αναγνώρισης και πιστοποίησης των αεροσκαφών και των συστημάτων τους και βεβαίως ε, ε, θα επεκταθεί η συμφωνία και όσον αφορά τους κινητήρες αλλά και όσον αφορά και τα υπόλοιπα αεροναυτικά προϊόντα και τα εξαρτήματα. Πιστεύω και θα ήθελα να απευθυνθώ και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ, πιστεύω ότι θα πρέπει και στο μέλλον να δούμε με ποιο τρόπο ε, θα ενημερώνεται έγκαιρα το Κοινοβούλιο για όλες τις περαιτέρω τροποποιήσεις που θα λάβουν χώρα αργότερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Ε, σχετικά με την ερώτηση που ακούσαμε για τον ρόλο του ε, Κοινοβουλίου, ερώτηση που ακούστηκε προηγουμένως από τον κύριο Ντεβάλε, ε, έχω μία έκθεση σχετικά με την δυνατότητα παρέμβασης του Κοινοβουλίου σε τέτοιες περιπτώσεις και βεβαίως τέτοιου είδους θέματα οπωσδήποτε θα μπουν στα, στις εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας. Θα πρέπει να ορίσουμε χρονικό όριο για τις τροπολογίες και θα πρέπει να διαβάσω λοιπόν τον, την προθεσμία είναι 4 Οκτωβρίου μετά για την Επιτροπή Μεταφορών 26-27 ε, και ψηφοφορία στην Ολομέλεια τον Νοέμβριο. Ορίστε, έκανα και το καθήκον μου σαν πρόεδρος. Πάρα πολύ ωραία. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι ανταλλαγή απόψεων με την ε, Επιτροπή σχετικά με την χρηματοδότηση των ΤΕΝ. Δεν ξέρω αν έχουν έρθει όλοι ε, και από την Επιτροπή. Τώρα διστάζω λίγο να χτυπήσω κουδούνι για διάλειμμα, αλλά μετά θα ξανάρθετε. Εν πάση περιπτώσει, 10 λεπτά. 10 λεπτά, γιατί μετά θα έχουμε σοβαρή συζήτηση για χρήματα. Να μην λείψει κανένας. 10 λεπτά λοιπόν διάλειμμα. Okay, don't go. We have the commission. Πού πάτε, μη φεύγετε. Ήρθε ο εκπρόσωπος Επιτροπής. Okay, colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Thank you. Είχαμε μιλήσει για δεκάλεπτο διάλειμμα, αλλά το ανακαλώ. Περνάμε στην ανταλλαγή απόψε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Η οριστική έκθεση της πεντεμεριλούς ομάδας των εμπειρογνωμόνων με επικεφαλή τον κύριο Σέτσι περιλαμβάνει συστάσεις για τις μελλοντικές δημοσιονομικές ανάγκες και το, τη γενική διάρθρωση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Προσκαλέσαμε τον κύριο Πακέ για να σας παρουσιάσει την έκβαση των συζητήσεων και τα πορίσματα της έκθεσης αυτής. είχαμε προσκαλέσει και τους προέδρους των ε, Επιτροπών Προπολογισμών, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, αλλά συμπίπτει δικός, ε, δυστυχώς η συνεδρίασή μας με τις δικές τους. Πάντως εγώ, που επειδή είμαι καλός άνθρωπος και επειδή διαπνέαμε από πνεύμα συνεργασίας, τους προσκάλεσα παρόλα αυτά. Και θα είναι και ευκαιρία να ακούσουμε όλοι της ε, θέσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτό το κεφαλαιόδε ζήτημα που είναι η χρηματοδότηση των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Γιατί κύριε Πακέ όλοι μπορούμε να κάνουμε ε, γραμμές ε, σε χάρτη, αλλά αν δεν έχουμε τα απαραίτητα κονδύλια θα μείνουν οι γραμμές στα χαρτιά και δεν θα περάσει, δεν θα γίνει τίποτα στην πράξη. Σας στοιχειωμένο μου φαίνεται αυτό το κοινοβούλιο. Κύριε Πάκη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής και των άλλων Επιτροπών και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου ξαναδίνετε για να σας παρουσιάσω την κατάσταση σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της πολιτικής για τα διευρωπαϊκά δικτύα μεταφορών. Να πω δύο λόγια διαδικαστικά καταρχήν, για να ενημερώσω και τους ευρωβουλευτές και Κατόπιν θα εμείνω στις ε, βασικές συστάσεις και πορίσματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Ετοιμάσαμε και κάποιες διαφάνειες, αλλά προτιμώ να τις μοιράσω γιατί είναι πολλές. Άλλωστε έχετε και την ε, έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Πριν από λίγους μήνες έγινε η διάσκεψη για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών στη Σαραγώσα και η δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε στόχο έχει να υποστηρίξει και να τροφοδοτήσει τη συζήτηση περί μεθοδολογίας για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. 15 Σεπτεμβρίου έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι δημόσιες ε, διαβουλεύσεις Έχουμε λάβει 220 230 προτάσει από διάφορα σώματα, Ινστιτούτα, Σωματεία κτλ. Ήταν ευρία η βάση αυτή τη δημόσιας διαβούλευση. Επεξεργαζόμαστε τώρα όλε αυτέ τι συνεισφορέ και θα καταρτήσουμε έκθεση που θα υποβάλουμε μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Η έκθεση δεν θα περιλαμβάνει μόνο πληροφορίε για την δημόσια αυτή διαβούλευση, αλλά όπω είπε και ο Επίτροπο Κάλλα στη Σαραγώσα, η έκθεση αυτή θα τελειοποιήσει ουσιαστικά την μέθοδο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δίκτυο των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και με το Κοινοβούλιο και να διατρανώσουμε αυτή τη συνένεση που δημιουργήσαμε με διαφανή τρόπο αλλά και με μία καλή και στιβαρή μεθοδολογία με συμμετοχή και συνεργασία με τα κράτη-μέλη, το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Έχουν απομείνει και κάποια κρεμή θέματα και για το βασικό δίκτυο και για τα υπόλοιπα, για το Core Network. Θα πρέπει να δούμε καταρχήν ποιοι είναι οι βασικοί κόμβοι. Φυσικά είπαμε 27 πρωτεύουσε για να έχουμε ευρία κάλυψη σε όλη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης τα βασικά λιμάνια θα συμμετέχουν στο δίκτυο και τα σημαντικά σημεία εισόδου στα ανατολικά σύνορα, αλλά θα πρέπει όλα αυτά να μπουν στο χάρτη και να αποφασιστούν και τα λιμάνια. Θα έχουμε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Λιμένων και φυσικά συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Μετά την ολοκλήρωση του βασικού δικτύου θα πρέπει να αποκρισταλώσουμε τι απόψει μα για το θέμα αυτό, χάρη και στη δημόσια διαβούλευση που έγινε. Επίση, θα πρέπει να προσδιορίσουμε τα βασικά οικονομικά κέντρα, τα οποία θα συνδέει αυτό το βασικό δίκτυο. Και επίση θα αξιοποιήσουμε το έργο τη Γενική Διεύθυνση ε, Περιφερειών και τη Διεύθυνση για την Εδαφική Συνοχή. Και έχουμε και την ΕΣΠΟΝ, θα την γνωρίζετε. Όλα αυτά θα μα βοηθήσουν Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν τα βασικά οικονομικά κέντρα που δεν είναι πάντα σωστά κατανεμημένα, διανεμημένα μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουμε λοιπόν συνεισφορές και των κρατών μελών και των ενδιαφερομένων για να τελειοποιήσουμε αυτό το θέμα. Επίσης και οι ροές της κυκλοφορίας μας ενδιαφέρουν, γιατί δεν θέλουμε να χαράξουμε μόνο κάποιες γραμμές στο χάρτη, αλλά να στηριχθούμε στις υπάρχουσες υποδομές, να δούμε πού βρίσκονται οι βασικοί σύνδεσμοι, αλλά να εντοπίσουμε και τις στενοπούς. Δηλαδή, πού υπάρχει κυκλοφορία και συμφόρηση σε ό,τι αφορά τις υποδομές, να κάνουμε προβλέψεις για την κυκλοφορία, να δούμε την πυκνότητα της κυκλοφορίας κτλ. Η όλη προσέγγιση για το βασικό δίκτυο, το Core Network, θα στηριχθεί στην προσπάθεια προσδιορισμού της ε, ε, μεγαλύτερης δυνατής προστιθέμενης αξίας ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα επικεντρωθούμε και σε προγράμματα ή συγκεκριμένα τμήματά τους που θα εντοπίσουμε στην εφαρμοστική φάση. Θα επανέλθω σε αυτό αργότερα όταν σας μιλήσω για τη στρατηγική χρηματοδότηση. Πάντως, το Core Network θα χρησιμοποιήσει την υπάρχουσα υποδομή, αξιοποιώντα την καλύτερη, με καλύτερη διασύνδεση των μέσων μεταφορά, με τα συστήματα διαχείριση μεταφορών και κυκλοφορία, μεγιστοποίηση τη δυνατότητά του και σε ορισμένε περιπτώσει τα νέα κυρίω κρατημέλη θα κατασκευαστούν και νέα τμήματα υποδομών. Ένα άλλο σημείο που γίνεται πλέον αρκετά κατανοητό και προέκυψε σαφώς από τη Σαραγώσα είναι ότι το Core Network θα είναι προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω αλλά θα έχει και ε, ε, θα έχει χαρακτήρα επιτακτικό. Δηλαδή, θα πρέπει να εφαρμόζεται και εγκαίρως και σωστά. Για το Core Network, αυτό το βασικό δίκτυο, είχαμε συνεργασία και με τα κρατημέλη, αλλά πολύ στενή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση MOVE, Γενική Διεύθυνση Regio και ιδιαίτερα με τα κράτη-μέλη που γνωρίζουν καλύτερα την κατάσταση των υποδομών στις χώρες τους. Αλλά είχαμε συνεργασία και με τους συναδέλφους από την εκτελεστική υπηρεσία για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Την Πέμπτη θα έχουμε συνάντηση στην, Επιτροπή, στην Διευθύνουσα Επιτροπή των ΤΕΝΤΗ και εκεί θα γίνει μια αντίστροφη τελειοποίηση, από κάτω προς τα πάνω δηλαδή, και με τα Comprehensive Network Layer θα στηριχτούμε στα υπάρχοντα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Θέλουμε τα κράτη-μέλη να εξυγχρονίσουν τις βάσεις τους για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Επίσης έχουμε ευρεία τέτοια δίκτυα διευρωπαϊκά, αλλά υπάρχουν πολλά κενά που θα πρέπει να πληρωθούν. Τα comprehensive network είναι σημαντικό τμήμα της ε, όλης διαδικασίας και τίποτα από το βασικό δίκτυο δεν μπορεί να υλοποιηθεί αν δεν στηρίζεται σε υπάρχουσα υποδομή και το πλαίσιο των ε, ευρύτερων δικτύων. Και επίσης θα πρέπει να εξασφαλιστεί η λειτουργία πρόσβασης στο βασικό δίκτυο. Άλλωστε τα ευρύτερα δίκτυα αποτελούν τη βάση πολιτικών, της πολιτικής για την Ευρωβινιέτα για παράδειγμα. Το έργο αυτό συνεχίζεται και ευελπιστούμε ότι θα δημιουργήσουμε μια σφαιρική εικόνα για το τι μορφή θα έχει το Comprehensive Network, αυτό το ευρύτερο δίκτυο. Θα πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ βασικού δικτύου και ευρύτερου δικτύου. Το ευρύτερο δίκτυο, το Comprehensive Network, είναι από κάτω προς τα πάνω, ενώ το βασικό δίκτυο, Core Network, είναι από πάνω προς τα κάτω. Το ευρύτερο δίκτυο είναι ε, μεικτό. Καλύπτει λιμένες, αερολιμένες, ιστορικές πλωτές οδούς κτλ. Και θέλουμε και ένα νέο στρώμα που θα παρτίζεται από τα συστήματα συνδέσμου που έχουν χαρακτήρα συνδυασμένων μεταφορών ώστε στο Comprehensive Network, στο ευρύτερο αυτό δίκτυο, να έχουμε συγκεκριμένη υλική υποδομή, ώστε να εξασφαλίσουμε την ένταξη του Core Network, που θα είναι συνδυασμένων μεταφορών. Και μια άλλη διαφορά είναι το Core Network είναι υποχρεωτικό, ενώ το Comprehensive Network είναι ενδεικτικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φάση της κατάρτισης των κατευθυντηρίων γραμμών. Αν ρίξετε μια ματιά στον προγραμματισμό και στη χρηματοδότηση, βλέπετε ότι το κοινό του σημείο είναι η εφαρμογή. Και ένας από τους λόγους που ζητήσαμε αναθεώρηση της πολιτικής διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και επειδή ενδιαφέρθηκε και το Κοινοβούλιο γι' αυτό, είναι προκειμένου να γεφυρωθεί αυτό το εφαρμοστικό χάσμα που διαπιστώνουμε. Γιατί υπάρχει αυτό το χάσμα της εφαρμογής. Καταρχήν, η πολιτική διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών είναι υπερβολικά φιλόδοξη και μερικές φορές ε, δεν μπορούσε να παρακολουθήσει την σχετικά ισχυρή χρηματοδότηση. Αλλά υπάρχει πρόβλημα και με το συντονισμό. Το συντονισμό μεταξύ των κρατών μέλων, το συντονισμό μεταξύ των διαφόρων πηγών χρηματοδότησης, ακόμη και εντός του κοινοτικού προϋπολογισμού και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε μικρές συνιστώσεις συστατικά υποδομών που αναπτύσσονται σε ένα διάδρομο ασυντόνιστα όμως μεταξύ τους και χωρίς να αξιοποιούν συνέργειες μεταξύ τους. Και δεν μιλούμε μόνο για διασυνοριακά ζητήματα. Ακόμη και σε, στο ίδιο κρατος υπάρχουν προβλήματα έλλειψης συντονισμού. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε διαφάνεια, θα πρέπει να αποφύγουμε σόρευση κονδυλίων, τήρηση της διαδικασίας, Πάντως, μερικές φορές οι διάφορες συνιστώσεις ε, λειτουργούν εκ παραλλήλου και δεν αξιοποιούνται οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων και επεμβάσεων. Και έρχομαι τώρα στην προσέγγιση της χρηματοδότησης. Ο Επίτροπος Κάλλας στην ακρόασή του, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έγγραφο διαβούλευσης του Μαΐου, επικεντρώθηκαν στην ανάγκη μεγαλύτερης ολοκλήρωσης, για να μην πω συγχώνευσης των διαφόρων μηχανισμών στήριξης. Αυτό ήταν ο στόχος μας. Και αυτή τη στιγμή εντατικοποιήθηκε το έργο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Γενικές Διευθύνσεις Regio και MOVE, ώστε το Core Network στο πλαίσιο προγραμματισμού να επικεντρωθεί σε συγκεκριμένα προγράμματα με προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία και μετά να έχουμε εφαρμοστικούς μηχανισμούς που θα τη χάνουν στενού συντονισμού ώστε στο μέλλον να αξιοποιούνται οι συνέργειες μεταξύ τους. Αυτά στα λόγια, αλλά και στα έργα, αν δείτε τον προπολογισμό του TNT, του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, γίνεται με τη βάση ε, πρόσκληση και υποβολή προσφορών επιλέγουμε διάφορα προγράμματα που προτείνουν τα κράτη-μέλη. Εμείς επιλέγουμε φυσικά τα καλύτερα από αυτά που μας προτείνουν, γιατί σε μερικές περιπτώσεις έχουμε περισσότερη ζήτηση από ό,τι προϋπολογισμό, από ό,τι διαθέσιμα κονδύλια. Η πολιτική συνοχή και η περιφερειακή πολιτική λειτουργούν με βάση κάποια προγραμματικά έγγραφα, οπότε η απόφαση για το ποιο πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί λαμβάνεται από τα κράτη-μέλη κυρίως με εξέταση φυσικά και συναπόφαση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά η απόφαση είναι κυρίως εθνική. Και στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, εκεί έχουμε περιπτωσιολογική ανάλυση των προγραμμάτων. Και με τέτοια λεπτομεριακή ανάλυση λαμβάνονται οι αποφάσεις δανειοδοσίας. Αυτά είναι τα βασικά εργαλεία στήριξης ε, και του κοινοτικού προϋπολογισμού ή της ΕΤΕ. Βέβαια εδώ ισχύουν πολλές διαφορετικές διαδικασίες απόφασης. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να εξασφαλιστεί συντονισμός μεταξύ των διαφόρων τμήματων, προγραμμάτων που βρίσκονται στον ίδιο διάδρομο. Εξού και ανάγκη για πιο ολοκληρωμένο σχέδιο, όπως φάνηκε και στο έγγραφο διαβούλευση που υποβάλαμε πριν τη Σαραγώσα. Οι δύο βασικοί μηχανισμοί θα είναι το βασικό δίκτυο, το Core Network, που θα προβλέπει τις νομικές υποχρεώσεις, έχει επιτακτικό χαρακτήρα και θα είναι τα προγράμματα που θα υποστηριχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο αφενός και αφετέρου. Στη συνεργασία με τους συναδέλφους Γενικής Διεύθυνσης Ρέτζιο θα καταλήξουμε σε ένα μηχανισμό προγραμματισμού ή ενιαίο ή ολοκληρωμένο. Θα δούμε. Πάντως υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον προκειμένου να εντοπίσουμε κάποια προγράμματα στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής και της περιφερειακής πολιτικής. Με βάση αυτό μπορούν να γίνουν και με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Και θα δούμε και το πώς θα δρομολογήσουμε τη συνεργασία με την ΕΤΕ. Ας περάσουμε τώρα πέρα από το, από το αρχικό πρόγραμμα και ας προχωρήσουμε λίγο σε περισσότερες λεπτομέρειες. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε ε, συστήσει μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που δουλεύει υπό την ε, προεδρία του συντονιστού Κάρλος Κιάκη με μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από μια σειρά ακαδημαϊκών και εκπροσώπων ιδιωτικών τραπεζών. Νομίζω ότι στην έκθεση αναφέρεται ο λόγος ε, για τον οποίο ενδιαφέρεται η Γενική Διεύθυνση μου να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, για τα επόμενα βήματα τα οποία προτίθεται να πάρει και επίσης ότι δεν πρέπει να περιοριστούμε σε συγκεκριμένα προγράμματα για δημιουργία συγκεκριμένων υποδομών, αλλά θα πρέπει να δούμε τις υποδομές σαν ένα σύνολο του ευρύτερου τομέα των μεταφορών. Να δούμε δηλαδή και τη δημιουργία νέων υποδομών, αλλά και την ε, συντήρηση των υποδομών αυτών και επομένως ε, η χρηματοδοτική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει υπόψη σε όλα τα στοιχεία αυτά. Στην έκθεση επίσης αναφέρονται ότι οι επενδύσεις ε, στον τομέα των μεταφορών εξακολουθούν να παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, εξακολουθούν βεβαίως να έχουν μεγάλο μακροοικονομικό αντίκτυπο στις μεταφορές και οι υποδομές αλλά και οι επενδύσεις στα συστήματα μεταφορών γενικότερα και, στην... και πρέπει να πω επίσης ότι τα λεγόμενα και αναφερόμενα στην έκθεση ευθυγραμμίζονται με την στρατηγική 2020, με τους στόχους για ανάπτυξη ε, σε άμεσο αλλά και μεσοπρόθεσμο και, και μακροπρόθεσμο συγγνώμη, ε, ορίζοντα. Πέρα από την δήλωση αυτή και την ανάλυση, ε, στην έκθεση γίνεται αναφορά σε τρεις περιοχές πρώτη περιοχή διερεύνησης ε, δυνατότητες ε, ε, του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού καθώς επίσης και διασύνδεσης μεταξύ του ευρωπαϊκού και των εθνικών προϋπολογισμών. Δεύτερη περιοχή διερεύνησης είναι πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, τα, τα, τα κέρδη των μεταφορών σε νέες επενδύσεις και τρίτον πώς μπορούμε να βελτιώσουμε ή να αναπτύξουμε εργαλεία τα οποία ε, θα βοηθήσουν την χρηματοδότηση των projects. Αυτή, αυτές οι τρεις περιοχές διερεύνησης θα πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστούν ε, από κοινού. Δηλαδή, ε, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει ε, ένα κατά κάποιο τρόπο tour de table, ένας γύρος τραπέζι για εξέβρεση ε, της χρηματοδότησης ε, των ε, projects, αλλά επίσης το κατά πόσον ο κύριος χρηματοδότηση είναι είτε ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός είτε οι εθνικοί προϋπολογισμή θα μας οδηγήσει σε, ένα, σε μια ενδεχόμενη ενδυνάμωση από τη μία ή την άλλη πλευρά. Οι εμπειρογνώμονες βεβαίως και ήταν αναμενόμενο προσπάθησαν να δουν τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζει ε, το Ταμείο Συνοχής σε την όλη διαδικασία και προφανώς ε, σε αυτήν την ε, περίπτωση φαίνεται να υπάρξει κάποια διάσταση μεταξύ των διευρωπαϊκών δικτύων και του Ταμείου Συνοχής. Είναι γεγονός βεβαίως ότι όλου αυτού του είδους τα προγράμματα μπορεί να έχουν σημαντικότατο αντίκτυπο σε τοπικό ή ε, σε περιφερειακό επίπεδο και ε, επομένως ε, η τριβή προκύπτει κυρίως από τον τρόπο μορφή διακυβέρνησης, δηλαδή ποιος είναι επικεφαλής και λιγότερο από την ίδια την ουσία των προγραμμάτων. Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό αφορά και την καινοτομία αφορά επομένως τον προπολογισμό για την έρευνα ε, στον τομέα των μεταφορών, την εξέβρεση ε, διαφορετικών πηγών ε, χρηματοδότησης για κάθε είδους μεταφορές, μπορεί να είναι αστικές μεταφορές, μπορεί να είναι εναλλακτικέ, μορφέ ή οτιδήποτε. Η δεύτερη διάσταση είναι η διάδραση ανάμεσα στο τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο και βεβαίως ε, εδώ γίνεται συζήτηση για το Core Network. Η συζήτηση επίσης γίνεται και όσον αφορά το, τα ποσοστά συγχρηματοδότησης και ε, πρέπει να βρούμε ποιο ε, είναι το, το ποσοστό το οποίο είναι ιδεοδέστερο και πλέον προσήκον έτσι ώστε να κινητοποιηθούν και οι ευρωπαϊκοί πόροι και τέλος βεβαίως και η διαδικασία της, των πολιτικών επιλογής. Ε, όσον αφορά τον τρίτο πυλώνα που ανέφερα, εδώ ε, μπορεί να υπάρξει μια διάσταση ε, απόψεων. Εν πάση περιπτώσει όμως θα πρέπει να γίνει, γίνεται ήδη η συζήτηση αυτή και στο Συμβούλιο. Το κύριο επιχείρημα είναι ότι ο τομέας των μεταφορών ε, αφορά μεγάλα δημοσιονομικά έσοδα για τον ε, προϋπολογισμό και επομένως ε, εάν κάνουμε ορθή χρήση των οικονομικών στοιχείων οδηγούμεθα σε ασφαλή συμπεράσματα. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να ασκηθεί πίεση στους εθνικούς προϋπολογισμούς και αυτό είναι πάντα ένα πολύ δύσκολο θέμα και εν πάση περιπτώσει Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποια θα είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά αυτό το δεύτερο κομμάτι των συμπερασμάτων ε, των εμπειρογνωμόνων. Αλλά ε, πέρα από το earmarking των ε, πόρων, νομίζω ότι η όλη συζήτηση για την χρηματοδότηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε, μια, ένα διαφορετικό ταμείο, Ευρωπαϊκό Ταμείο Μεταφορών και μια διαφορετική ε, μορφή. Θα δούμε ε, με ποιο τρόπο μπορούν να χρησιμοποιηθούν, να, να εξευρεθούν έσοδα, μπορεί να ε, δημιουργηθεί αυτή η ευρωβιγέτα ή οτιδήποτε άλλο. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά τα οποία προτείνουν οι εμπειρογνώμονες είναι πολύ ενδιαφέροντα, αλλά ακόμα θα πρέπει να το συζητήσουμε. Τρίτο σκέλος, τρίτο στατικό είναι η χρηματοδότηση. Εκεί δίνεται μια πολύ, γίνεται μια πολύ καλή ανάλυση των περιορισμών και των δεσμεύσεων που ε, υφίστανται αυτή τη στιγμή, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ε, γίνεται συγκεκριμένη αναφορά ε, και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στο ενδεχόμενο κυκλοφορίας ευρωομολόγων. Σε γενικές γραμμές η ανάλυση που κάνουν για την αγορά και την κατάσταση αγοράς είναι περίπου ίδια ε, με αυτή που είχαμε κάνει και εμείς. Βεβαίως το πρόβλημα είναι ε, πώς είναι δυνατόν να διασφαλιστεί είτε η ε, κυκλοφορία ευρωομολόγων είτε άλλου είδους τίτλων που όμως θα είναι αρκετά ελκυστικοί έτσι ώστε να τραβήξουν, να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών στο παρελθόν και αυτό είναι βεβαίως τεχνικής φύσεως ε, στοιχείο και ελπίζω να μην με ρωτήσετε πολλά πάνω σε αυτό γιατί δεν είναι ο τομέας μου, δεν το ξέρω. Ε, εν πάση περιπτώσει ε, παλιότερα ε, υπήρχε, υπήρχαν τα χέγγια για αυτού του είδους της εκδόσης τίτλων. Λόγω της οικονομικής κρίσης δεν υπάρχει πλέον η ασφάλεια που υπήρχε παλιά και επομένως Ε, και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η χρηματοδότηση γιατί έχουμε και μεγάλη μείωση των εισόδων από 115 σε περίπου 60 ε, εκατομμύρια. Εν πάση περιπτώσει στην ε, έκθεση που μας απασχολεί γίνονται πολλές προτάσεις και όσον αφορά κάποιες εναλλακτικέ λύσεις και όσον αφορά το Ταμείο Μαργαρίτα και όσον αφορά σχετικά δηλαδή με άλλες άλλες ε, διευκολύσεις ε, έτσι ώστε να μπορέσουν να ε, γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις και για να κινητοποιηθεί όσο γίνεται μεγαλύτερος αριθμός πόρων και συμπληρωματικών και η συμπληρωματικών πόρων. Τα ομόλογα, από όσο ξέρω, ήταν και μία παλιά ιδέα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, αλλά εδώ η έννοια είναι διαφορετική, ε, δηλαδή να, γίνουν, να εκδοθούν ε, ομόλογα έτσι ώστε να, να, χρηματοδοτηθεί η ανάληψη κινδύνου. Αυτά ήθελα να σας πω, συγγνώμη που μακρηγόρησα. Ε, πρέπει να ε, βεβαιωθούμε ότι και η Επιτροπή σας ε, παραμένει με ενεργό ρόλο στην όλη διαδικασία. Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε όσον αφορά το πλαίσιο και οπωσδήποτε θα συνεχίσουμε και να σας δίνουμε την απαραίτητη πληροφόρηση όπως κάναμε και μέχρι τώρα άλλωστε. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο τώρα στους συντονιστές των ομάδων και θα αρχίσω τον κύριο Γκρός από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την δήλωση, την ανακοίνωση, όσων μπορεί να ανακοινώσει εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών. Κάποια κριτική ας μην την πάρουν προσωπικά, αλλά ως όργανο. Πολλά από όσα ακούσαμε εδώ είναι ξαναειδωμένα πράγματα. Και όχι μόνο τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, αλλά και τα τελευταία χρόνια τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Η δική μου ανησυχία είναι, όταν εξετάζω δηλαδή την διαδικασία που ακολουθείτε, είναι ότι αποφεύγουν τα ουσιώδη θέματα, εγκύπτοντας σε πράγματα τα οποία είναι γνωστά και χίλιες φορές αναλυμένα. Ίσως υπάρχουν τρία βασικά θέματα το εξή. Τι πρέπει να κάνουμε, δεύτερο, ποιο αποφασίζει και τρίτο, ποιο χρηματοδοτεί, ποιο πληρώνει. Το πρώτο το έχουμε απαντήσει ξανά και ξανά το πρώτο ερώτημα. Το μόνο που ίσως είναι νέο στοιχείο εν είναι κάτι που θα το αναμέναμε πιο πριν, δηλαδή ένα συντονιστικό έργο ανάμεσα στα όσα γίνονται στο περιφερειακό επίπεδο με ευρωπαϊκά χρήματα. Το δεύτερο και τρίτο ερωτήματα είναι στην ουσία θέματα που δεν αφαίρονται τόσο πολύ στην χρηματοδότηση, αλλά στην πολιτική βούληση. Να γίνει κάτι ή να μην γίνει. Τα όσα μέχρι τώρα ήδη έχουν συζητηθεί, χρειάζεται βέβαια να εξεταστούν. Αλλά αν, υπάρχει, αν υπάρξει αύριο η πολιτική βούληση να χρησιμοποιηθούν οι πόροι που βρίσκονται σε ορισμένα ταμεία για να αναπτυχθεί ένα κόνσεπτ κινητικότητας στην Ευρώπη, δεν θα χρειαστούν πολλές αναλύσεις, θα χρειαστούν στην βάση της πολιτικής αυτής λίγες φράσεις μόνο που να... ότι αυτοί οι πόροι διατίθενται για το τάδε έργο. Και αυτό είναι όλο. Σε ό,τι αφορά την χρήση τώρα των πόρων, όπως είπατε ήδη, νομίζω ότι αφενός οφείλουμε να αναμένουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε στη διάθεσή μας λιγότερα χρήματα, άρα πρέπει να τα δαπανίσουμε αποτελεσματικότερα. Δεύτερον, οι πηγές για τα χρήματα αυτά, είτε υπάρξουν νέε είτε είναι οι ίδιες οι παλές, θα πρέπει να τις εκμεταλλευτούμε καλύτερα, εάν δεν διασφαλίσουμε εδώ από την Επιτροπή Μεταφορών, αλλά και σε συνεργασία με το Συμβούλιο, ότι τα έσοδα, τα μελλοντικά έσοδα που θα προκύψουν να χρησιμοποιηθούν και στον τομέα της κινητικότητας ανεξαρτήτως του τρόπου, είτε πρόκειται για earmarking, είτε πρόκειται για ανάληψη υποχρεώσεων, να γίνουν με τρόπο τόσο ελκυστικό ώστε οι χώρες να θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά, να τα βάλουν στην συγχρηματοδότηση, δηλαδή να δοθούν κίνητρα. Τέλος πάντων, ανεξαρτήτως του τρόπου, Εάν δεν τα καταφέρουμε να γίνει αυτό, τότε ας λησμονήσουμε ολόκληρη την στάση, ε, ολόκληρη τη συζήτηση μάλλον της εσωτερικοποίησης του κόστους. Γιατί τότε έχει χαθεί η ευκαιρία. Αν οι χώρες δεν συμφωνήσουν στο Συμβούλιο ότι καλούνται να κάνουν επενδύσεις στον τομέα αυτό και να χρησιμοποιήσουν και τις νέες ενδεχομένως πηγές εσόδων που θα βρουν για τον σκοπό αυτό, τότε δεν έχει και νόημα. Οι αναλύσεις λοιπόν που κάνω τώρα μου δίνουν το εξής αποτέλεσμα. είναι ερωτήματος. Πότε θα μπορούμε να αναμένουμε τις σημαντικές, ουσιώδεις πολιτικές αποφάσεις, αυτά τα τρία σημαντικά ερωτήματα από την Κομισιόν αλλά και από το Συμβούλιο. Και με ποιον τρόπο μπορούμε να αναμένουμε μια ξεκάθαρη τοποθέτηση. Διότι δεν νομίζω ότι οι διάφορες αναλύσεις που γίνονται θα οδηγήσουν εν τέλει στην απάντηση των θεμελιωδών αυτών ερωτημάτων. Σωστές οι προετοιμασίες, αλλά οι προετοιμασίες αυτές θα ακυρωθούν εν τέλει εάν δεν απαντηθούν οι δύο σημαντικές, οι τρεις πάντων σημαντικές ερωτήσεις. Δηλαδή, πρώτον, ποιος θα αποφασίσει αύριο, μπορούν μόνες τους οι χώρες μέλη που διαχειρίζονται τα χρήματα της Ένωσης, είτε θα είναι το Κοινοβούλιο ή το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν που θα δώσουν κάποιες κατευθύνσεις. Δεύτερον, πώς θα συνδυάσουμε τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας στο επίπεδο της Ένωσης. Ευχαριστώ κύριε Γκρός. Αλκαντράουι από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. είχαμε μιλήσει και πριν τη συνεδρίαση με τον κύριο Κρός. Και εγώ την ίδια γνώμη έχω για το θέμα αυτό. Και το κεντρικό θέμα είναι τι ισχύ θα έχει αυτή η έκθεση των εμπειρογνωμόνων που βρήθη προτάσεων. Το θέμα είναι πώς θα τις αξιοποιήσουμε. Θα εστερνιστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα πορίσματα αυτής της έκθεσης. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε ορισμένα μόνο σημεία, γιατί δεν έχουμε γενναιόδωρο προϋπολογισμό. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε ορισμένα θέματα. Καταρχήν, θέλουμε περισσότερη διαφάνεια. Περιμένουμε προσδιορισμό των κριτηρίων. Πρώτα θα πρέπει να προσδιορίσουμε τα κριτήρια, ώστε να μπορέσουμε κατόπιν να προτείνουμε κάτι πιο συγκεκριμένο. Επίσης, πολλές προτάσεις κατατέθηκαν, ώστε τα πενιχρά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας να τα αφιερώσουμε στα 10 σημαντικότερα σημεία στις 10 στενοπούς που έχουμε στην Ευρώπη. Και με βάση αυτή τη φιλοδοξία της κατάρτισης των στενοπών θα πρέπει να χαράξουμε τις 10 προτεραιότητές μας είχαμε πει ότι αν θέλουμε ως κοινοβούλιο να υλοποιήσουμε κάτι σημαντικό θα πρέπει να δούμε τι μέσα διαθέτουμε για τα διάφορα σχέδια και, και φυσικά να εξετάσουμε τα διασυνοριακά τμήματα. Επίσης θα πρέπει να βελτιώσουμε και το συντονισμό να ενισχύσουμε τις αρχές συντονισμού. Και όλα αυτά να γίνουν αποτελεσματικά, αλλά θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις. Αν θέλουμε να συμφωνήσουμε και για τα μέσα και για το συντονισμό, θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να ενδώσουν σε ορισμένα ζητήματα. <coughs> Γιατί μιλούμε για τα χρηματοδοτικά μέσα Μιλάμε για την Ευρωβινιέτα. Συμφωνούν τα κράτη-μέλη θα μας δημιουργήσουν προβλήματα. Θα συμφωνήσουν οι χώρες μέλη με τις προτάσεις, γιατί δεν θα είναι ανεφόρον αυτή η ευρωπαϊκή ενίσχυση. Θα πρέπει απέναντι στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουμε και τα ενάβσματα και τις απειλές και το καρότο και το ραβδί για να μπορέσουμε να έχουμε ένα αυτό πολιτικό αποτέλεσμα. Και η πρώτη προϋπόθεση είναι η ίδια Επιτροπή να υποβάλει μια όσο πιο φιλόδοξη πρόταση γίνεται και μακρόπνοη. Αν το τολμήσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βρει το Κοινοβούλιο στο πλευρό της. Δυστυχώς όμως δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο από δημοσιονομική άποψη, γιατί τον προϋπολογισμό τον καθορίζουν και τα κράτη-μέλη που ζητούν επενδύσεις σε ένα δυναμικό δίκτυο μεταφορών. Στα λόγια, αλλά στα έργα δεν λαμβάνω συγκεκριμένες δράσεις. Η κυρία Μάισνερ. Ο κύριος Γκρός είπε ήδη ότι αυτά τα πράγματα είναι ξαναειδωμένα και δίκιο θα έχει. Εγώ είμαι ε, καινούρια εδώ και δεν τα ξέρω τόσο καλά. Οι μεταφορές είναι η ραχοκαλιά της ενιαίας αγορά και επομένω είναι απαραίτητε. Τα γνωρίζουμε αυτά. Επίση είναι λίγα τα χρήματα που έχουν οι μεταφορέ στη διάθεσή του ώστε να βελτιωθούν πραγματικά οι υποδομέ που χρειάζεται να βελτιωθούν. Συμβαίνει λοιπόν ξανά και ξανά να βλέπουμε ότι τα λεφτά που έχουν οι χώρε στη διάθεσή του πρέπει να δαπανηθούν με τον αποτελεσματικότερο τρόπο. Κύριε Πακέ, είπατε και μου φάνηκε λίγο αστείο όπω το είπατε ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τι χρηματοδοτικές δυνατότητε. Εγώ νομίζω ότι μάλλον το ξεχάσαν αυτό. Είπαν, είπε ο καθένα τι ήθελε για να ικανοποιηθούν όλε οι χώρε μέλη. Τα συζητήσαμε αυτά και στη Σαραγώσα τη Ισπανία. Και τελικά δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Εν πάση περιπτώσει, από τα πολλά που ε, υπάρχουν, εμεί είπαμε ότι πρέπει ορισμένα να προκριθούν. Να δούμε ποια είναι τα πιο σημαντικά και μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Μιλήσατε και για την υψηλότερη δυνατή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Πραγματικά, πού βρίσκεται αυτή, σε οικονομικά κέντρα ή, όπως θεωρήσαμε εμείς, σε διαμεθωρια... διαμεθοριακά έργα. Διότι οι χώρες συνήθως σχεδιάζουν μέχρι τα σύνορά τους. Ο σχεδιασμός τους παίρνει μέχρι τα σύνορά τους. Και εκεί θα έπρεπε να παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Σαραγώσα λοιπόν σκεφτήκαμε πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν και βέβαια πρέπει όντω να προχωρήσουμε. Είναι βέβαια δύσκολο γιατί σημαίνει να δοθεί προτεραιότητα σε ορισμένα έργα προτεραιότητα. Κάτι το οποίο θα πονέσει ορισμένου. Κανέναν δεν θέλουμε να πονέσουμε, αλλά είναι αναγκαίο. Θα παραμείνει λοιπόν δύσκολη επιλογή. Αυτό είναι σαφώς για σαφές για μένα. Δεν έχουμε ούτε και ταμείο ειδικό για τις ε, υποδομές μεταφορών, κάτι που ήθελε ο Επιτρόπος, αλλά δεν συμφώνησαν οι κυβερνήσεις. Είπαν οι κυβερνήσεις για ποιο λόγο να φτιάξουμε και άλλο ταμείο, ας τα αφήσουμε όλα στο περιφερειακό ταμείο. Ίσως μια μερική λύση να είναι η Ευρωβινιέτα σε συνδυασμό με το earmarking, που ίσως μπορεί να δώσει κίνητρο στις χώρες μέλη να εισπράττουν τέλη από κάποιες ε, οδούς, κάποιους αυτοκινητοδρόμους ή σχετικές διόδους και να τα χρησιμοποιούν μετά αυτά για χρηματοδοτήσεις. Και η ερώτησή μου είναι τι γίνεται εν τέλει με την επιλογή των προτεραιοτήτων, την προτεραιότητα που θα δοθεί στις προτεραιότητες δηλαδή, με ποιο τρόπο θα αντιμετωπιστεί αυτό. Ευχαριστώ. Κυρία Λίχτενμπέργκερ, από τους Πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξέτασα προσεκτικά τα έγγραφα. Πίνακες όπως τούτος εδώ που σας δείχνω είναι πραγματικά πολύ κοπιαστικό να αναγνωστούν και δύσκολο να ερμηνευτούν. Και εν τέλει αυτά που ε, δείχνει ο πίνακας, τι να πω τώρα, ε, είναι ωραία και πολύ χρωμή αλλά αυτονόητα δεν είναι. Ίσως να οφείλεται στο ιδιαίτερο στυλ της Κομισιόν, αλλά θα σπάσουν τα κεφάλια τους οι πολίτες για να καταλάβουν τι ακριβώς θέλουμε. Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται και οι προκαταλήψεις κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι είναι πολύ απομακρυσμένοι από τους πολίτες. Σας παρακαλώ λοιπόν, φτιάχτε κάπως ε, διαγράμματα και πίνακες που να εξηγούν καλύτερα τα πράγματα. Τώρα για την ουσία. Πρώτα, μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Εδώ αμέσως σκέφτομαι την Ευρωβινιέτα. Η πρόταση για το earmarking, εγώ πάντα την έχω υποστηρίξει και μου αρέσει. Μου φαίνεται και σωστή. Αλλά να μην πάνε τα χρήματα όλα αυτά πάλι στην κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, ώστε να υπονομευτούν οι στόχοι που έχουμε διθέσει και αυτός ο, αυτή η πολυτροπική ε, προσέγγιση πρέπει να διατηρηθεί. Τώρα, βρισκόμαστε εν μέση διαδικασία λήψης αποφάσεων ε, από πλευρά Συμβουλίου για την Ευρωβινιέτα. Όταν λέτε σήμερα ότι οι χώρες εκείνες μέλη οι οποίες επιθυμούν να εισαγάγουν την Ευρωβινιέτα θα πρέπει ευθύ αμέσω να διοχετεύουν τα εισπρατώμενα χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μη γνωρίζοντας πού θα χρησιμοποιηθούν, ε, τότε θα, θα κερδίσει το λόμπι των φορτηγατζίδων, διότι ποτέ, πουθενά δεν πρόκειται να εισαχθεί αυτό το ευρωσήμα ή η ευρωβινιέτα. Μόνο εάν γίνει υποχρεωτικά, τότε καλά. Τι γίνεται τώρα. Ευρωβινιέτα, ίσως οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί, και τα χρήματα θα τα βάζουν σε ένα καλάθι που δεν θα γνωρίζουν από εκεί πέρα που θα πάνε. Αυτό πολιτικά είναι ανεφάρμοστο. Δεν πρόκειται να γίνει. Ερχόμαστε λοιπόν και προσφέρουμε μια κηδεία τρίτης τάξεως σε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο αρχικά πρόγραμμα. Εάν είναι από την αρχή ξεκάθαρο ότι τα λεφτά κάπου θα χαθούν όπου καμία χώρα μέρος θα γνωρίζει πού θα πάνε, αυτό λοιπόν μπορείτε να ξεχάσετε ότι θα προχωρήσει. Είναι ξεκάθαρα ένα από τα παραδείγματα εκείνα τα οποία είναι σχέδια ωραία στα χαρτιά που δεν πρόκειται ποτέ να υλοποιηθούν στην πράξη. Το άλλο που δεν μπορώ να καταλάβω είναι αυτή η διατηρούμενη αισιοδοξία σε αυτή την υπόθεση της ε, σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Υπάρχει και έγγραφο της ίδιας της Κομισιόν που λέει ότι αυτή η σύμπραξη δεν λειτουργεί στις μακροπρόθεσμες ε, στρατηγικές, στις, μακροπρόθεσμα, στις μακροπρόθεσμες χρηματοδοτήσεις οι οποίες θα αποσβεστούν σε 50 χρόνια. Λειτουργεί ίσως η σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα μοναχά σε βαχυπρόθεσμα έργα. Ένα ερώτημα. Ελπίζω όταν λέτε την καλύτερη χρήση των υφιστάμενων υποδομών, ελπίζω να μην εννοείται άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας την νύχτα των φορτηγών αυτοκινήτων ή αλλαγή των ορίων βάρους και διαστάσεων, διότι θα προκληθεί σύγκρουση και νομίζω επίσης ότι για παράδειγμα αυτές οι εντάσεις ανάμεσα στο Ταμείο Συνοχής και στα διευρωπαϊκά δικτύα. Αυτά τα πράγματα είχαν αποφασίσει κάποιοι πρωθυπουργοί τότε που σήμερα δεν έχουν πλέον τίποτα, κανένα λόγο στην ε, πολιτική ζωή των χωρών. Άρα βρεθείτε λίγο καλύτερα με τα δύο σας πόδια να πατάτε στη, στο έδαφος της ε, σημερινής ε, πολιτική πραγματικότητα. Και όταν λέτε ότι θα πρέπει να γίνουν υποχρεωτικά, σε μια χώρα μέλο και δεν εννοώ μοναχά τι νέε χώρε μέλη, αλλά και ορισμένε από τις παλαιέ, σε μια χώρα μέλο, όπου δεν υπάρχουν χρήματα, ε, πώς θα τους αναγκάσετε. Όπου δεν υπάρχουν χρήματα, χάνει και ο βασιλιάς το δίκιο του, λέει μια παλιά γερμανική παροιμία. Πώς λοιπόν θα το εφαρμόσετε. Στη θεωρία ωραία είναι αυτά που λέτε, αλλά στην πράξη μάλλον μου φαίνεται ότι θα δυσκολευτείτε. Και τέλος χαίρομαι που αξιολογείτε περισσότερο τα λιμάνια. Ευχαριστώ κύριε Λίχτενπέργκερ. Και εσύ και εμείς ε, στα αγγλικά λέμε αν δεν έχετε λεφτά μηδέν θα πάρετε. Της κυρίας Μάισνερ Τώρα, από την εκλογική της περιφέρεια, έχουμε μια ομάδα επισκεπτών. Καλώς ήλθατε όλοι στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Δεν ξέρω αν και στο πρώτο μισό ήταν εδώ η ε, μισή από την ομάδα επισκεπτών. Εν πάση περιπτώσει, καλώς ώρες μας σε όλες και όλους σας. Και ελπίζω να σας φανεί ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σήμερα ήταν πολύ σημαντική μέρα για την κυρία Μάισνερ, γιατί υπερψηφίσαμε το πρωί την πρώτη της έκθεση στην Επιτροπή. Και περνάμε στις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Παρακαλώ να μην ξεπεράσετε το τρίλεπτο για να προλάβουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί φαντάζομαι κομμένη την ανάσα της περιμένετε. Ο κύριος Κάντσαν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον ε, κύριο Πακέ παρκέ. Και ε, μακαρίζω και την συνάδελφο που έχει αυτό το περιβόητο πίνακα, έγχρωμο μάλιστα. Εγώ ούτε ασπρόμαυρο δεν τον έχω. Εν πάση περιπτώσει, συμφωνώ με αυτά που είπε ο συντονιστής μου, ο συνάδελφος Γκρός, και μέσα στα τρία λεπτά που μου δώσατε θα επιχειρηματολογήσω σχετικά με την ανάγκη ελάχιστης προγραμμα... ελάχιστου προγραμματισμού και υλοποίησης και σεβασμού των χρονοδιαγραμμάτων. Ο προγραμματισμός βεβαίως είναι σωστός, αλλά τα πράγματα έχουν πολύ αλλάξει με τους νέους αυτοκινητοδρόμους, με τις, με τις νέες λεωφόρους κυκλοφορίας της Ευρώπης. Έχει αλλάξει πολύ η εικόνα. Η υλοποίηση τώρα. Σχετικά με την υλοποίηση, νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε μέθοδο πλέον και να προσανατολιστούμε προς τη δημιουργία ενός ταμείου, που δεν θα είναι όμως ένα ταμείο συνοχής ή ένα ταμείο παρόμοιο με αυτά που έχουμε σήμερα και που βλέπουμε ότι δίνουν στην ουσία υποτροφίες ή δίνουν χρήματα χωρίς ε, καμία ελπίδα επιστροφής, αλλά να ε, εξερευνήσουμε άλλες οδούς που τελικά θα αναπτύξουν και θα χρηματοδοτήσουν κάτι το οποίο είτε με κάποιο, είτε τέλος πάντων θα μας αποφέρει, θα αποφέρει κάποια χρήματα, είτε ε, θα μας δώσει κάποια επιστροφή ε, χρημάτων. Πιστεύω ότι εάν εμείς βάλουμε από τη μία μεριά την νομική βάση των λεωφόρων και από την άλλη την νομική βάση των ε, ταμείων, τότε μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο όργανο το οποίο πραγματικά θα μας βοηθήσει. Τώρα, πώς θα χρηματοδοτηθεί το ταμείο αυτό, με τι θα προοικοδοτηθεί αφενός με την εξοικονόμηση που θα έχουμε από άλλα ταμεία, μεταξύ αυτών και το Ταμείο Συνοχής. Δεύτερον, να είναι χρήματα τα οποία δεν θα τα δώσουμε θα τα χάσουμε, αλλά θα μπορέσουν να μας επιστρέψουν ε, κάποιο κέρδος. Τρίτον, θα πρέπει να προσπαθήσουμε μέσω την, ε, της Ευρωβινιέτας, μέσω της ε, διεθνούς, του διεθνούς ορισμού τιμών, ε, να ε, κάνουμε ε, μια καλή δουλειά έτσι ώστε να συνδυαστούν να συνδυαστούν τα κόστη των μεταφορών, τα οποία γνωρίζουμε ότι τώρα είναι πάρα πολύ ψηλά. Το έγγραφο των 5 ανοιχνεύει πολύ ορθά τις δυνατές οδούς. Αναφέρει δε κάπου τη δημιουργία ενός ταμείου που θα ελέγχεται ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από, το, ε, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και θα μπορέσει να ε, συνδυάσει τον, τον δημόσιο ε, με τον ιδιωτικό τομέα ε, και τις χρηματοδοτήσεις τους. Νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη σκέψη μας έτσι ώστε να δώσω σε όλους να καταλάβουν ότι μιλάμε πλέον για ένα ταμείο το οποίο θα είναι διαφορετικό, δεν θα είναι ε, σαν αυτό το ταμείο συνοχής ε, ή σαν οποιοδήποτε άλλο ταμείο. Θα είναι κατά κάποιο τρόπο μία λεωφόρος ε, η οποία μέσω συγκεκριμένων δανείων, μέσω της J, μέσω άλλων μέσων θα οδηγήσει σε ένα καλό αποτέλεσμα. Η κυρία Γιάννα Σέντερς. Ευχαριστώ. θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Πακέ για την παρουσίαση που μας έκανε, γιατί αυτό μας έλειπε ουσιαστικά για να ολοκληρώσουμε τη Γενική Επισκόπηση και το μεθοδολογικό σκέλος πριν αρχίσουμε τη μάχη, κατά κάποιο τρόπο. Συμφωνώ με τον κύριο Καντζάν. Πιστεύω ότι είναι απολύτως απαραίτητο, εν ώψη της συζήτησης που έχει ξεκινήσει για τον επόμενο πολίτη προϋπολογισμό, να λάβουμε υπόψη την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα ειδικό ταμείο μεταφορών, που θα πρέπει να είναι αυτόνομο. Και αν στι προηγούμενε δημοσιονομικέ προοπτικέ δώσαμε έμφαση στην έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη και πραγματοποιήσαμε ένα ποιοτικό άλμα, στι νέε δημοσιονομικέ προοπτικέ ήρθε η ώρα να δώσουμε έμφαση στην κινητικότητα, τι υποδομέ και την καινοτομία στι μεταφορέ. Αυτό θα πρέπει να είναι το πολιτικό μα μήνυμα για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Και υπάρχει και ένα άλλο τμήμα. Το θέμα της αξιολόγησης ε, της επίπτωσης που θα έχει ένας ανεπαρκής προϋπολογισμός για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Είδατε τι έγινε με την Ισλανδική Φεστιακή Τέφρα. Είδατε τι έγινε με την ε, απεργία στη Γαλλία ή την αυριανή απεργία στο Βέλγιο, αν δεν αποτραπεί δεν μπορούμε να έχουμε ένα μόνο μέσο. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τις οδικές μεταφορές με άλλα μέσα. Γι' αυτό θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποτιμήσει τον, την επίπτωση μιας ανεπάρκειας του προϋπολογισμού για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Στην έκθεση ΠΕΣ προτείναμε μέσω του Golden Rule να μετατρέψουμε το δημοσιονομικό έλλειμμα σε παραγωγικές επενδύσεις σε υποδομές. Και ο κύριος Κώστα πρότεινε το γαλλικό μοντέλο, αλλά τι ακριβώς εννοεί. Αυτό που είναι σημαντικό και μας το λένε και τα κράτη-μέλη, είναι ότι θα πρέπει να επενδύσουμε σε υποδομές χωρίς να τρέχει το κοντέρ του δημοσιονομικού ελλείμματος Ω κάτι αρνητικό μόνο. Να έχουμε και κάτι θετικό, που θα είναι οι επενδύση στι υποδομέ. Και να αξιολογήσουμε και τις επιπτώσεις ενό τέτοιου μέτρου. Αλλά και η διακυβέρνηση είναι σημαντικό θέμα. Δύνατη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπροσωπήσει τα κοινοτικά συμφέροντα ώστε να υποχρεώσει κατά κάποιο τρόπο τα κράτη-μέλη σε αυτή τη νέα φάση να συγχρηματοδοτήσουν τα προγράμματα που θα πρέπει να συγχρηματοδοτήσουν. Και σε ό,τι αφορά την Ευρωβινιέτα, θα ήθελα να ρωτήσω, μπορεί επικαλούμενοι το κοινοτικό συμφέρον να υποχρεώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα κράτη-μέλη να αφιερώσουν τμήματα κονδύλια στις μεταφορές. Εγώ κάνω ό,τι μπορώ στην Ισπανία, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί ισχύει ένας κανόνας που λέει ότι όλα θα πρέπει να πάνε στο Υπουργείο Οικονομίας. Υπάρχει το ενιαίο ταμείο. Δεν ξέρω αν μπορεί να μας βοηθήσει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και για τις επιχορηγήσεις, για τα μπόνους, υπάρχουν τέτοια προηγούμενα. Δηλαδή, κοινοτικέ πολιτικές να χρηματοδοτούνται από, από τα ομόλογα, συγγνώμη. Και είναι, θα ήταν ελκυστικά τέτοιου είδου ομόλογα αν κυκλοφορεί στην αγορά. Κύριε Μάλτερ, αν δεν με κοιτάτε θα χτυπάω πιο δυνατά το σφύρι. Περίμενα, περίμενα να με καλέσετε. Είμαι νέο μέλος στην Επιτροπή αυτή. Καταρχήν να δούμε το θέμα της χρηματοδότησης των προγραμμάτων. Έχουμε διάφορε ε, πηγέ χρηματοδότηση, το κοινοτικό προπολογισμό, του εθνικού προπολογισμού, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τι συμπράξει δημοσίου και ιδιωτικού φορέα. Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για το μερίδιο των διαφόρων αυτών πηγών χρηματοδότηση. Για να δούμε στι χείουσε δημοσιονομικέ προοπτικές ποια ήταν η συμμετοχή των διαφόρων πηγών χρηματοδότηση, Με ενδιαφέρουν τέτοια στοιχεία. Και για το μέλλον δεν έχω και πολλές ελπίδες για το μελλοντικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί σε όλες τις χώρες γίνονται περικοπές στους εθνικούς προϋπολογισμούς, οπότε δεν έχω και πολλή αισιοδοξία για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τον αυξήσουμε. Θα μπορούσαμε όμως να δώσουμε περισσότερες εγγυήσεις στην ΕΤΕ. Αυτό γίνεται ήδη για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Υπάρχει μια αντίστοιχη δημοσιονομική γραμμή και υπάρχει και αποθεματικό με εγγύηση των εθνικών κυβερνήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πληροφορίες για το τι απο... ποιο είναι το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα αυτών των εγγύσεων. Γιατί έχουμε 100 εκατομμύρια εγγύσεις στον προϋπολογισμό. Πόσα δάνεια μπορούμε να δώσουμε με τέτοιου είδους εγγύηση. Και τέλος, πάλι κοιτάω τον πρόεδρο. Ποιο είναι το ποιο ποσοστό των οδών στην Ευρώπη χρηματοδοτούνται από συμπράξεις ιδιωτικών και κρατικών φορέων. Και πώς μπορούμε τέτοιου είδους ε, δάνεια να τα χρηματοδοτήσουμε από ιδιωτικούς επενδυτές, ιδιώτες επενδυτές. Έχει παραδείγματα τέτοια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, κύριε Μάλντερ. Συγχαρητήρια. Κάτι που θα είναι δύσκολο να τηρηθεί. Τρία λεπτά, κύριος Κράμαρ. και ε, άλλη παροιμία εδώ εισαγωγικών εμεί οι Γερμανοί που λέμε είναι άμα δεν ξέρω τι να κάνω φτιάχνω μια επιτροπή αλλά και η Κομισιόν νομίζω κάπως έτσι το βλέπει το πράγμα δεν λειτουργούν τα πράγματα αυτά δεν λειτουργεί ο σχεδιασμό των ε, διευρωπαϊκών δικτύων γιατί βλέπουμε και στο τοπικό και στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο παντού τα ίδια πράγματα. Πώς θα τα αλλάξουμε εμείς. Για παράδειγμα, όταν έπεσε στο τείχος του Βερολίνου αντιμετωπίσαμε το ε, δίλημα θα φτιάξουμε 5 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ε, υπόγειο σιδηρόδρομο που θα χρειαζόταν 30 χρόνια ή θα, φτιάχναμε 5 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομο μέσα σε 3 χρόνια. Και επέλεξε το δεύτερο το Βερολίνο. Και άλλα παρόμοια έργα μπορώ να σας αναφέρω. Ούτε ξέρουμε και πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα αυτά. Επομένως για τα επόμενα 10 χρόνια θα απορροφήσουν το 70% των διατηθειμένων κονδυλίων. Το τρίτο τώρα στην Ευρώπη από τα 30 διευρωπαϊκά δίκτυα που στην ουσία είναι ένα συνονθήλευμα ε, εθνικών εγωισμών. Έχουμε μονάχα το τούνελ Μπρένερ, το ναυτοκινητό του Τουρίνου, Μεσίνα και άλλο ένα. Αυτά τα τέσσερα λοιπόν έργα, είτε διπλασιαστεί ο προπολογισμό του, είναι έτοιμα σε 30 χρόνια κατά το 40, 50, 60 ή 70% δεν παίζει κανένα ρόλο, διότι κανένα δεν αζήσει μέχρι τότε για να τα δει. Άρα πρέπει να συνδυάσουμε την έγκριση ενός έργου με την υποχρέωση συγχρηματοδότησης. Εάν στη Γερμανία ήταν υποχρεωμένες οι ομόσπονδες χώρες ή οι δήμοι και οι κοινότητες να προβλέψουν χρηματοδότηση για τα επόμενα 10 χρόνια σε ένα έργο που εγκρίνει η Ομοσπονδική Κυβέρνηση, όλα αυτά τα έργα θα μειώνονταν κατά πολύ σε αριθμό και θα είχαν τη δυνατότητα να δημιουργηθούν. Ε, Φέρνω το παράδειγμα της Ιταλίας, από τις πιο σημαντικές και πλούσιες οικονομικά ε, ε, χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τρία που ανέφερα, το τούνελ του Μπρένερο, η Μεσίνα κτλ. Και όλοι γνωρίζουν ότι οι Ιταλοί δεν πρόκειται ποτέ να τα καταφέρουν να φτιάξουν αυτά τα πράγματα. Ποτέ. Δεν είναι δυνατόν. Παρ' όλα αυτά δίνονται ξανά και ξανά χρήματα. Άλλο παράδειγμα. Στην Ισπανία, αυτοκινητόδρομο, ο οποίο κατασκευάζεται με κοινοτική χρηματοδότηση. Και είναι σχεδόν άδειο. διότι είναι τόσο ακριβά τα διόδια, τα οποία ωστόσο χρηματοδοτήσαμε με 85% εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε τα φορτικά αυτοκίνητα πηγαίνουν από τους εθνικούς δρόμους. Το ίδιο συμβαίνει και αλλού. Όσο λοιπόν δεν αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα, μπορούμε να συζητούμε για καινούργια ταμεία, για παραπάνω χρήματα, ό,τι θέλετε μπορούμε να συζητούμε, αλλά είναι περιτά. Πρέπει να εξετάσουμε τα αίτια. Ωραία είναι τα ευχολόγια, αλλά είναι για τα Χριστούγεννα οι πολιτικοί, όπω είμαστε εμεί, όριμοι άντρε και γυναίκε, θα ότι τα ευχολόγια δεν αποδίδουν τίποτα. Τρεμόσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μου αρκεί ένα λεπτό για να ευχαριστήσω τον κύριο Πακέ που ήρθε στο Κοινοβούλιο να μας παρουσιάσει τα πόρισματα της έκθεσης και να πω ότι η πρότασή του ότι τα προγράμματα που θα επιλέξουμε θα πρέπει να έχουν αυξημένη προστιθέμενη αξία είναι πολύ σωστή. θα πρέπει προηγουμένως να γίνει μία ανάλυση κόστους-οφέλους για να προσδιοριστούν τα μακροοικονομικά ωφέλη των διαφόρων διαδρόμων. Αυτό θα μας βοηθούσε να κάνουμε πιο σωστές επιλογές και να έχουμε περισσότερα ωφέλη και πλούτο. Και συμφωνώ με την κυρία Μάισνερ ότι θα πρέπει να κάνουμε μια επιλογή και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Αυτό το λάθος κάναμε στους αυτοκινητοδρομούς που κατασκευάσαμε στην Ισπανία, που δεν μπορέσαμε μακροοικονομικά ωφέλη να δρέψουμε από τα έργα αυτά εξαιτία της ε, κακής επιλογής της θέσης τους. Επίσης έχουμε το πρόβλημα των στενοπών σε ορισμένες χώρες ή μεταξύ κάποιων χωρών μελών. Και ας μην ξεχνούμε ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουμε και την, ε, ολοκληρω... την ενιαία αγορά. Από το 19ο αιώνα ε, ζητούν οι καταλανικές εταιρείες ε, μια απελευθέρωση και υπάρχουν προβλήματα ακόμη και στην ίδια τη χώρα. Ευχαριστώ. Θα είμαι και εγώ σύντομο. Ο δόκτωρ Πακέ που εξήγησε λεπτομερώς την διαδικασία μπορεί να πει και λίγα λόγια για την σημερινή κατάσταση του προϋπολογισμού. Τα 103 δισεκατομμύρια, τα 130 μάλλον, τα 130, 130 δισεκατομμύρια που έχουμε στη διάθεσή μας από αυτά προβλέπονται λίγα για την χρηματοδότηση των μεταφορών και γνωρίζουμε και ποιες είναι και τα χρονικά περιθώρια. Γι' αυτό η αφετηρία που εξηγεί ο κ. Πακέ λέει ότι οι χώρες μέλη πρέπει να αξιολογήσουν ποια έσοδα προέρχονται από τον τομέα των μεταφορών μέχρι τώρα διόδια για βαριά φορτηγά αυτοκίνητα. Μιλήσαμε και για Γαλιλαίο και τηλεματική. Πρέπει να βάλουν κάτω όλα τα έσοδα και αυτά να θεωρηθούν ως συγχρηματοδότηση για τέτοια έργα των διευρωπαϊκών δικτύων. Όταν μιλάμε για ρέγγι και για τα ταμεία των υποδομών, προβλέπονται εκεί συγκεκριμένα ποσοστά των πόρων για τις υποδομές. Και από τα 130 δισεκατομμύρια το 40% προβλέπεται γι' αυτό, για αυτούς τους σκοπούς. Και είναι σημαντική η προσανατολάς διεύρυνση πάλι εν προκειμένου. Αν θέλουμε να έχουμε την δυνατότητα να υλοποιήσουμε σε κάποιο ορατό μέλλον τα διευρωπαϊκά δίκτυα και για τη Γερμανία, επειδή αναφέρθηκε η χώρα μου πριν. Μόνο για τα τρένα υπάρχει χρηματοδότηση ευρωπαϊκών δικτύων, ενώ υπάρχουν και άλλα πράγματα όπως ο Ρήνος ή η Βόρεια Θάλασσα που θα μπορούσαν... Μα όλα είναι για το σιδηρόδρομο. Μην έρχεστε αντίθετη τώρα με την δική σας την πολιτική και να λέτε ότι δεν είναι δυνατόν να ε, επενδύονται χρήματα σε κατασκευή σιδηροδρομικών σταθμών. Θυμίζω την Στουτγάρδη 21. Από... Υποτίθεται ότι θα φτιάξουμε το σιδηρόδρομο που θα διέρχεται όλη την, σχεδόν όλες τις κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες. Ευχαριστώ κύριε Κούν. Θα κατάλαβα. Ε, επισκέπτεσαι ότι ε, πήγαινε σημαντικές περιφερειακές εκλογές στη Γερμανία. Πριν ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Πακέ για να απαντήσει, να κάνω κι εγώ σύντομα σχόλια. Συμφωνώ με τον κύριο Μιλντερ για, τη χρηματοδότηση. Να βρούμε τρόπους να χρηματοδοτήσουμε τα διάφορα προγράμματα. Αναφέρθηκε η πρόταση Μπαρόζο για τα ευρωομόλογα. Εγώ έχω επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά τις συμπράξεις ε, ιδιωτικού και κρατικού φορέα τέτοιου είδους συμπράξεις είναι θεωρητικά καλές. Στην πράξη όμως κολλάνε γιατί το, το κέρδος ε, το δρέπεται ο ιδιωτικός φορέας και τον κίνδυνο τον αναλαμβάνει ο κρατικός. Αν υπάρχει όντως ε, πραγματική σύμπραξη ιδιωτικού και κρατικού φορέα θα πρέπει όχι μόνο το κέρδος ε, να είναι κοινό αλλά και οι υποχρεώσεις να μοιράζονται αν μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε σωστά, εντάξει, αλλά Όπω είπε και ο κύριο Πέρντερ, επειδή θα υπάρξουν περικοπές στου εθνικούς προπολογισμού, θα δούμε πω εμεί θα αυξήσουμε τα κονδύλια για τα προγράμματα αυτά. Και τέλο, ε, η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Ακούσατε κύριε Πακέ από πολλού ευρωβουλευτέ ότι είναι σημαντικό το θέμα τη ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Παρά είναι μακροσκελής ο κατάλογος των προτεραιοτήτων. Θα πρέπει να θυσιάσουμε ορισμένες από αυτές να παραιτηθούμε από ορισμένε. Και σίγουρα κάποια κράτη θα δυσαρεστηθούν για την απομάκρυνση κάποιων προγραμμάτων, αλλά το Ταμείο είναι μείον, γι' αυτό και θα πρέπει να είμαστε πιο μετριοπαθείς. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια σωστή ιεράρχηση των προτεραιοτήτων. Κατά τη γνώμη μου, αν επιζητούμε ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και πραγματικά διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, τότε θα πρέπει να ασχοληθούμε κυρίως με το διασυνοριακό τους χαρακτήρα. Και ακόμη και η υψηλή ταχύτητα, οι μεγάλες ταχύτητες σταματά στα σύνορα γιατί δεν τηρούν όλες τις υποχρεώσεις στα κράτη-μέλη. Και αυτό θα είναι και η λιδιαλήθος για την πρόοδο. Αν έχουμε τρένα υψηλής ταχύτητας Περπινιάν, Βαρκελόνης, τότε είναι θα μπορούμε να πούμε ότι κάναμε κάποια πρόοδο. Κύριε Πακέ, Σύντομα παρακαλώ. Ήταν βέβαια πληθώρα οι ερωτήσει που υπευλήθησαν, αλλά αν μπορείτε να είστε σύντομος και να απαντήσετε όσο πιο συνοπτικά γίνεται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής. Να είναι γεγονός ότι προηγουμένως κάλυψα πολύ έδαφος, αλλά ε, ενδεχομένω ε, μπορώ να κάνω και μερικά σχόλια επιπλέον απαντώντας ερωτήσεις που ε, τέθησαν. Δεν είμαι σίγουρος αν θα πρέπει να ξεκινήσω από το τέλο με τη συμπράξη ιδιωτικού και κρατικού φορέα. Ε, ο σκεπτικισμός όσον αφορά αυτές τις ε, ε, συμπράξεις βεβαίω είναι πάρα πολύ λογικέ, αλλά γνωρίζουμε πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει ένα, μια πραγματική καλή σύμπραξη ιδιωτικού κρατικού ε, και οι παράμετροι είναι πάρα πολλές, δηλαδή οι δυνατότητες που έχει η κάθε πλευρά, ε, από ποια περιφέρεια, από ποια χώρα. Ε, επομένως, οι παράμετροι είναι πάρα πολλές έτσι ώστε να γίνει μια σωστή σύμπραξη. Και κύριε Μούλτορ, αν έπρεπε να δώσω έναν... Κατανοούμε τώρα όσον αφορά τον δημο, τον, ε, τους προϋπολογισμούς αυτών των ε, συμπράξεων. Ε, πρέπει να πω ότι χρηματοδοτούνται 70% από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% από τα κράτη-μέλη και υπάρχουν και κάποια ε, και, ένα ε, υπόλοιπο το οποίο δεν αφορά χρηματοδοτήσεις ε, άμεσης αλλά προς επιστροφή. Όσον αφορά τώρα τα στοιχεία αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο, στη σχετική μας έκθεση όπου αναφέρονται και όλες οι προτεραιότητες. Τώρα, η χρηματοδότηση των projects και όχι απαραίτητα οι συμπράξεις λοιπόν η χρηματοδότηση των project σαν ένα σκέλος της διαδικασίας ολοκλήρωσης ε, οπωσδήποτε παραμένει ένα σημείο ανοιχτό, είναι ένα θέμα το οποίο ε, αντιμετωπίζουν ε, οι εμπειρογνώμονες και βεβαίως μας απασχολεί. Μας απασχολεί δε το να δούμε εάν μπορούμε σε ολόκληρη την λεωφόρο και σε διασυνοριακό επίπεδο να κρατήσουμε κάποιες βασικές και απαράλλακτες αρχές. Ενδεχομένως ένα τμήμα λοιπόν της διαδικασίας να χρειάζεται ένα ομόλογο του είδους που ανέφερα προηγουμένως ή ε, σε κάποιο άλλο σημείο μια επιπλέον χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τη χώρα μέλη. Ε, μέλος. Εν πάση περιπτώσει, ε, το θέμα είναι αν δημιουργήσουμε μία λεωφόρο θα πρέπει να δούμε ποια είναι η δυνατή χρηματοδότηση, ποια είναι η δυνατότητα ολοκλήρωσης των project κτλ. και επομένως έτσι να καθορίσουμε και την γενικότερη ευρύτερη στρατηγική μας όσον αφορά την χρηματοδότηση με οποιαδήποτε μορφή. Νομίζω ότι ε, καλύφθηκαν όλα τα στοιχεία. Αυτό που παραμένει ακόμα να πω είναι ότι θα πρέπει να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο ε, θα γίνουμε αποτελεσματικότεροι και πώς είναι, ε, θα καταστεί δυνατόν να παραγάγουμε αυτήν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για το πρώτο, πώς θα είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Έχει συζητηθεί πολλές φορές το θέμα αυτό. Ε, και το έχουμε πει και με εσά. Το ζήτημα είναι να χρησιμοποιήσουμε την υπάρχουσα υποδομή ε, και να γίνει μέσω ε, καλής διαχείρισης των ροών να γίνει πιο αποτελεσματική η χρήση. Καλύτερη λοιπόν αποτελεσματικότερη χρήση των υποδομών και βεβαίως να βρούμε τρόπους με τους οποίους θα βελτιώσουμε την βάση γνώσεων, έτσι ώστε να ξέρουμε ποια είναι τα κομμάτια τα οποία χρειάζονται επιπλέον, ε, επιπλέον χρηματοδότηση. Ένας τρόπος είναι να πούμε τι χρειάζεται η λεωφόρος από το Βερολίνο στο Παλέρμο και ένας άλλος τρόπος είναι να δούμε τα μεμονωμένα τμήματα επί των οποίων μπορούμε να επιφέρουμε βελτιώσεις. Το βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μια σωστή βάση γνώσης έτσι ώστε να μπορούμε να απομονώσουμε με τις ε, ε, ανάγκες ε, και να βρίσκουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Αυτό που δεν ανέφερα προηγουμένως είναι το θέμα των προτύπων. Δηλαδή, χρειαζόμαστε τρένα υψηλής ταχύτητας παντού, χρειαζόμαστε μια ενιαία λύση παντού. Αυτό επίσης είναι μια ξεχωριστή συζήτηση σχετικά με τις προτεραιότητες και την αποτελεσματικότητα των επιλεγόμενων προτεραιοτήτων. Απομένως καλύτερη στοχοθέτηση των αναγκών, λαμβάνοντα υπόψη τις ε, υπάρχουσες δυνατότητες και τις μελλοντικές προοπτικές. Κατά αυτή την έννοια πιστεύω ότι οι σοβαρότερες προτεραιότητες είναι αυτές οι οποίες δίνουν την μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία ε, και ε, μπορεί να ακολουθηθεί είτε μια διασυνοριακή λογική είτε μια ή μια διαδικασία εχμής. Ε, Βεβαίω και όσον αφορά τις ε, διατροπικές μεταφορές πολύ περιθώριο υπάρχει ακόμα για συζήτηση. Η διατροπικότητα μπορεί ε, να ωφελήσει, μπορεί να μας, ε, ε, αν τη μαζί με τα πρότυπα, μπορεί να μας οδηγήσει σε πάρα πολύ καλές, σε πάρα καλά αποτελέσματα. Επομένως, μεγάλη προτεραιότητα δίνουμε στην διασύνδεση των τρόπων μεταφοράς. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Αλλά βεβαίω σε κάθε περίπτωση χρειαζόμαστε και ε, καλή πληροφόρηση για όλα τα projects. Επόμενη ερώτηση είναι η εξής. Με βάση όλα αυτά μπορούμε να επιτύχουμε με τα κράτη-μέλη και μέσω και του Συμβουλίου και του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί ε, να φτάσουμε στη δημιουργία ενός ε, ε, ε, πυρηνικού δικτύου, γιατί βεβαίως το, ο κίνδυνος είναι να βάλουμε σε αυτό το πυρηνικό δίκτυο πολλά ε, ε, πράγματα και να το βαρύνουμε. Ε, αυτό που μας ενδιαφέρει να δημιουργήσουμε λοιπόν αυτόν τον πυρήνα που θα αποτελεί ένα παράδειγμα για κάθε επίπεδο οικονομικό, αποτελεσματικότητας κτλ. Και να επικεντρωθούμε σε αυτό και για μία ακόμα φορά λέω ότι ο ρόλος αυτού του πυρηνικού δικτύου είναι να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τα επόμενα 15-20 χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι χρειάζεται απολύτως νέα υποδομή για όλη, για όλη την Ευρώπη και παντού. Αυτή είναι μια διαλεκτική η οποία έχει ήδη ξεκινήσει με τα κράτη-μέλη. Βεβαίως πολλή δουλειά έχουμε μπροστά μας. Ένα από τα κύρια μηνύματα της ε, Σαραγώσας ήταν ένα νέο πνεύμα. Δηλαδή ότι και η Κομισιόν και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ε, βγήκαν από την Σαραγώσα πεπισμένοι ότι πρέπει πρέπει να συνεχίσουμε, ε, ότι όμως χρειάζονται αμοιβέ δεσμεύσεις ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι με αυτά εν μέρη τουλάχιστον απαντώ στις ερωτήσεις σας. Μία τελευταία παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε, ε, σχετικά με την προσέγγιση διαλεοφόρων. Σαφώς υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου των Ευρωπαίων συντονιστών και ε, βεβαίως θα πρέπει με πιο συντονισμένο τρόπο να ε, ληφθούν οι αποφάσεις που θα φορούν τα χρηματοδοτικά μέσα. Και από αυτόν βεβαίως εργάζεται ο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Α, ναι, όσον αφορά την ε, Ευρωβινιέτ, κυρία Λίτνεμπεργκερ, όντως έχετε δίκιο Στην έκθεση όντως αναφέρεται ότι για να είναι ε, το earmarking αποτελεσματικό, ε, μάλλον δεν κάνει λόγο μόνο όμως για earmarking, ε, αναφέρεται σε διάφορους τρόπους χρήσης ε, των ε, χρημάτων από την Eurovignet, δηλαδή ε, σε εθνικό επίπεδο να πηγαίνουν σε ένα ταμείο τα χρήματα για την Ευρωβινιέτα, από την Ευρωβινιέτα μάλλον, και ένα τμήμα να πηγαίνει σε ένα ευρύτερο ταμείο. Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανάγκη για earmarking, αυτό τουλάχιστον αναφέρει η έκθεση και σίγουρα είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητηθούν επιπλέον. Ε, εκτός και αν δεν κατάλαβα καλά αυτό που είπατε. Πολύ σύντομα. Η δική μου ερώτηση ήταν διαφορετική, λέει η κυρία Λίχτενμπέργκερ. Το σύστημα αυτό, δηλαδή της δυνατότητας να υπάρχει ένα ποσοστό υπέρ του Ταμείου Μεταφορών με την έννοια ότι είναι οικειοθελές αυτό θα καταστρέψει όμως ε, το ευρωσήμα, την ευρωβινιέτα. Ή προβλέπετε ότι ενδεχομένως μπορεί κάποτε να γίνει υποχρεωτικό. Αυτό είναι για μένα το ερώτημα. Νομίζω ότι κατάλαβα σωστά την ερώτησή σας και απάντησα τι λέει η έκθεση των εμπειρογνωμόνων. Ε, γιατί λόγω της θέσης μου είναι δύσκολο να απαντήσω απευθείας ε, εξ ονόματος του οργάνου μου στην ερώτησή σας. Σας ευχαριστούμε κύριε Παρκέ. Περιμένουμε ανυπόμονα την ολοκλήρωση της γραμμής Βαρκελόνη-Περπινιάν. Γίνομαι κουραστικός με την επανάληψη. Σας ευχαριστώ για τη συζήτηση. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημέρης της διάταξης, σε σχέδιο έκθεσης Κράμερ για την πολιτική ανταγωνισμού του 2009. <coughs> Μάικλ, θα μας κάνεις παρακαλώ μια σύντομη εισαγωγή. Ταιριάζει και με τη συζήτηση που μόλις κάναμε, διότι υπήρχε αθέμητο συνταγωνισμό στην Ευρώπη. Παράδειγμα, έχουμε τα υποχρεωτικά διόδια των σιδηροδρόμων που ισχύει για κάθε μηχανή έλξεως ανεξαρτήτως εάν μεταφέρει εμπορεύματα ή ε, επιβάτες και έχετε από την άλλη μεριά οικειοθελώς ε, διόδια των αυτοκινητοδρόμων, δηλαδή αν θέλει κάποια χώρα μέρο θα επιβάλλει και μόνο για φορτηγά άνω των 12 ετών κτλ. Γιατί λοιπόν το κάναμε αυτό, διότι αναζητούσαμε και επιζητούσαμε τον θεμητό ανταγωνισμό. Έτσι λοιπόν δεν είχαμε θεμητό ανταγωνισμό μεταξύ των τρόπων μεταφοράς, ούτε όμως και γενικότερες μεταφορές. Γι' αυτό πρέπει να εξεταστεί όχι μονάχα αν υπάρχει ανταγωνισμός, πρέπει να ε, καταλαμβάνει και όλους τους τρόπους μεταφοράς και να μην εξετάζει μονάχα το χρήμα αλλά και γενικά τις ιδέες που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως, κυρίως την ανάγκη προστασίας του κλίματος, την αναχέτηση της αλλαγής αυτής, διότι εάν δεν τα εφαρμόσουμε αυτά δεν πρόκειται να αναχέτησουμε την αλλαγή του κλίματος και βεβαίως δεν είναι μονάχα το θέμα οικολογία και οικονομία, είναι και η κοινωνική διάσταση. Η διατήρηση των προδιαγραφών ε, χρόνου εργασίας, ασφάλειας κλπ, χρηματοδότηση των υποδομών, όλα αυτά λοιπόν θέλουμε να περιληφθούν, διότι υπάρχουν 30 δισεκατομμύρια ευρώ που πληρώνει κάθε χρόνο ο ε, Ευρωπαίος φορολογούμενος υπέρ των αεροπορικών εταιριών, διότι αυτές είναι απαλλαγμένες από φόρους καυσίμων κλπ. Αυτά πρέπει να τα πούμε, να τα γνωρίζει ο κόσμος. Αυτά που είπα στην αρχή λοιπόν, υποχρεωτικά διόδια στον σιδηρόδρομο ή και ο θελός στα αυτοκίνητα. Το ίδιο ισχύει και για τους επιβάτες. Για τα αεροπλάνα είπαμε αποζημίωση σε περίπτωση καθυστερήσεων από 5 ώρες και μετά ενώ για τα τρένα είπαμε από την πρώτη ώρα κιόλας 25%, τη δεύτερη ώρα 50%. Πάλι αυτό είναι αθέμητο σε βάρος του σιδηροδρόμου. Τώρα ήρθε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και μείωσε από τις 5 ώρες στις 2,5 ώρες για τα αεροπλάνα. Αυτό είναι ντροπή για μας. Εν πάση περιπτώσει τώρα, ανεξαρτήτως του αυτοκινήτου υπήρχε υποστήριξη από το δημόσιο τομέα. στηρίζοντας τους αυτοκινητοδρόμους που είναι αυτοί που με τη σειρά τους καταστρέφουν το κλίμα. Τώρα, ε, στην παράγραφο μου παριθμών 6 υπογραμμίζω την ανάγκη να αποφευθεί ο του ανταγωνισμός για να διατηρηθούν οι κοινωνικοί κανόνες και σε θέματα ασφαλείας και περιβάλλοντος. Μας είπαν τότε Καμιά φορά μας λένε οδηγοί φορτηγών αυτοκινήτων παίρνουν τηλέφωνο ε, από το κινητό τους τηλέφωνο και λένε οδηγώ ήδη 12 ώρες με αναγκάζει ο εργοδότης μου παρακαλώ σταματήστε με και ελέγξτε με το λένε οι ίδιοι τροχοί. χρειάζεται λοιπόν να εξεταστεί το θέμα αυτό δεν είναι δυνατόν μια επιχείρηση να εξαναγκάζει τους εργαζομένους της ε, να παραβιάζουν τον νόμο ώστε να υποφελείται η ίδια επιχείρηση Επίσης, πρέπει να εξετάσουμε τις ειδικές συνθήκες που ισχύουν και στις ενέργειες μεταφορές. Υπάρχουν περιφερειακά αεροδρόμια τα οποία ε, δεν ε, αποδίδουν μεταξύ Μάνχαιμ και Ζαρβρουκεν, για παράδειγμα, που είναι σε ξεχωριστές ομόσπονδες χώρες. Ας πούμε λοιπόν, λένε οι χώρες, χρειαζόμαστε 2.000 εισιτήρια από το Ζαρβρουκεν μέχρι το Βερολίνο. τα δίνουν αυτά. Κάνουν τρίκ λοιπόν, δίνοντας έτσι έμεσες επιδοτήσεις. Αυτά τα βλέπουμε, τα βλέπουμε και αλλού. Στην παράγραφο μου παριθμών 8 λέμε first time, first time, last time. Δεν μπορεί να υπάρχει κρατική ενισχύση για τις αερομεταφορές. Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία λέει ότι η επιδότηση αυτή μπορεί να γίνει άπαξ μόνο. Ξέρουμε ότι στην Ιταλία και στην Ελλάδα παραβιάστηκε κατ' επανάληψη η διάταξη αυτή. Και εδώ πρέπει λοιπόν να εφαρμοστούν και να τηρηθούν οι νομοθεσίες. Θεματοφύλακας των συνθήκων είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη στο πρώτο πακέτο τα είχαμε συζητήσει. Εννέα χρόνια μετά φτάνουμε στην ιδέα να τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά και να τα υλοποιήσουμε, να τα εφαρμόσουμε. Εδώ η αμοιβαιότητα επίσης Υπάρχουν χώρες οι οποίες τα πάνε μια χαρά στον ανταγωνισμό τους μέσα σε άλλες χώρες, αλλά δεν τον επιτρέπουν μέσα στη δική τους επικράτεια. Αυτό δεν το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Από το 2007 και μετά. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν χώρες οι οποίες δεν επιτρέπουν τον ανταγωνισμό στους σιδηροδρόμους στην επικράτειά τους. γνωρίζοντας ότι εν τέλει θα επιδοτηθούν. Και εδώ λοιπόν οφείλουμε να διδαχθούμε. Και στην αυσιπλοεία υπάρχουν οι μεγάλες κοινοπραξίες οι οποίες έχουν χωρίσει την αγορά σε κομμάτια. Δεν μπορεί κανείς να συζητεί καν περί ανταγωνισμού εδώ. Και εδώ πρέπει να, καταργηθεί, να καταργηθούν αυτές οι, αυτά τα εμπόδια. Στην τελευταία μου παραγραφή που δεν μπορούσα να τη βάλω στην έκθεσή μου αλλά τα είπα και πριν στην συζήτηση ότι καταργήθηκε ο φόρος ε, σε βάρος των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων στη Γαλλία, αλλά τώρα έχει επιβληθεί ένα τέλος τροχαίου υλικού, με το αποτέλεσμα ότι οι αλλοδαπές επιχειρήσεις να πληρώνουν το φόρο επιχειρήσεων στην χώρα τους, αλλά και να πληρώνουν και το τέλος τροχαίου υλικού στην Γαλλία. Ενώ οι ντόπιοι σιδηρόδρομοι τα περνάνε μια χαρά. Πρόκειται πάλι για θέμη του ανταγωνισμού και μέσα στην ευρωπαϊκή ενιαία αγορά. Δεν πρόλαβα να το γράψω στην εκθεσή μου αυτό, αλλά όπως είπε ο Ματίο Γκρός, θα υποβάλει ε, τροπολογία μαζί μου και θα το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη μου πρόταση. Αν έχετε συμπληρώσεις ή βελτιώσεις, πολύ ευχαρίστω να, να μου τις θέσετε υπόψη μου. Να συνεργαστούμε όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να μην μακρηγόρησα, αγαπητέ Πρόεδρε. Καθόλου ήσουν και εισηγητής. Ο κύριος Κούν από το ΕΛΚ. Δυστυχώς κολλείεται σήμερα ο κύριος Μπαχ που είναι ο εισηγητής μας για την υποβολή ερωτήσεων στις προτάσεις του κύριου Κράμερ για το δίκαιο ανταγωνισμού στον τομέα των μεταφορών. Σε πολλά πράγματα βρισκόμαστε σε συνένεση μαζί του, ίσως εκπλήξουμε τα υπόλοιπα μέλη τη Επιτροπής, γιατί έχουμε διαφορετικέ επιχειρηματολογίε ο κ. Κράμερ και εγώ συνήθω. Είναι σημαντικό βέβαια να προχωρήσουμε σε μια συνολική ενατένιση του προβλήματος. Για το, στην παράγραφο 2, για παράδειγμα, οι διαρθρώσεις των τιμών πρέπει να είναι απλές και διαφανείς. Γιατί συχνά ο πελάτης ή ο επιβάτης είτε στο σιδηρόδρομο, είτε στις εναέρειες μεταφορές, είτε στην αυσιπλοεία, είτε στη μεταφορά επιβατών. Στην ουσία είναι άοπλος απέναντι στην πολιτική διαμόρφωση των τιμών. Στην παράγραφο 3 είναι σημαντικό και εδώ να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει από τις χώρες μέλη να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Με ποιον τρόπο δηλαδή ορίζουν, καθορίζουν και διαρθρώνουν τις κρατικές ενισχύσεις τους. Αντί να πάμε και να λέμε ανακλάδο μεταφοράς ε, αν ο σιδηρόδρομος ε, λαμβάνει ενισχύσεις ή όχι, όπως είπατε κύριε Κράμερ ε, και είπατε για τη Γαλλία ότι ε, καταργεί τον φόρο ε, των γαλλικών σιδηροδρόμων αλλά βάζει ένα τέλος τροχαίου υλικού που πλήττει πλέον όλους. Αυτά είναι λοιπόν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, οι, οι, οποίες, οποίες στρεβλώσεις μάλλον εν τέλει μας παρεμποδίζουν από το να φτιάξουμε την ενιαία αγορά που όλοι επιθυμούμε. Λίγα λόγια για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες που είναι αρμοδιότητα ε, της ε, Επιτροπής Μεταφορών. Ο Σίμψον ως εισηγητής το έχει πει κατ' επανάληψη και το έχει αναλύσει. Θα πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, καθορίσει αυτή την καθολική υπηρεσία και του δημοσίου συμφέροντος και να την διευκρινίσει, να την, να την ορίσει δηλαδή σαφώς, να εξηγήσει πού βρίσκονται οι ασάφειες, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και ο ιδιωτικός τομέας, αλλά και να ανταποκρινόμαστε και στην βασική καθολική αυτή υποχρέωση που έχουμε, ώστε ο κάθε άνθρωπος δηλαδή να έχει το δικαίωμα να λαμβάνει την αλληλογραφία του στον τόπο διαμονής του. Για την παράγραφο 4, κύριε Κράμερ, αναφέρεστε μονάχα στο σιδηρόδρομο, αλλά στα προφορικά που είπατε, αναφερθήκατε και σε δικαιώματα επιβατών κλπ. Αυτό πρέπει να ισχύσει για όλους τους ε, φορείς μεταφορών. Κάτι που δεν προκύπτει από την γραπτή σας διατύπωση εδώ. Για την παράγραφο 5, δεν ξέρω αν την κατανοώ σωστά, πώς η ενίσχυση της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει επιπτώσει στην παγκόσμια αγορά. Γιατί δηλαδή το βάζετε αυτό εδώ να το βάλετε στην ανάλυση του τι ακριβώς είναι κρατική ενίσχυση. Δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποια παράγραφο, αλλά εκεί θα, μπορείτε, εκεί θα μπορέσετε να, να βάλετε την ιδέα αυτή. <clears throat> Κατά τα λοιπά μας ικανοποιεί η γνωμοδότηση. Αυτό το first time, last time, ίσως να το εκλαϊκεύσετε κάπως, ενώ την παράγραφο 8, να το εκλαϊκεύσετε κάπως το καταλάβουν περισσότεροι. Ευχαριστώ. Λάιχτφριντ, ευχαριστώ. Αντικαθιστώ την σκιώδη συγγήτρια κυρία Τικάου. Ε, υπάρχουν πολλά μικρόφωνα ανοιχτά και δεν ακούμε καλά τον ομιλούντα. Λοιπόν, για αυτά για την κριτική που θα πω δεν ευθύνεται ο εισηγητή. Θα πω τώρα ότι κατά βάση η τη εισηγητρία συμφωνεί με την πρόθεση του εισηγητού. Η μόνη ένσταση που ίσως έχει είναι ότι ενδεχομένως χρειάζεται μια καλύτερη κατανομή σε ό,τι αφορά τις ρυθμιστικές διατάξεις και τις διατάξεις περί ανταγωνισμού. Εγώ προσωπικά δεν το βρίσκω τόσο σημαντικό, αλλά η σκιώδη συγγήτρια θεωρεί ότι, για παράδειγμα, στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 4, οι ρυθμιστικές διατάξεις είναι λίγο υπερβολικές, όχι επί της ουσίας, αλλά για την παρούσα πρόταση και που από όσο ξέρω θα κατατεθούν κάποιες τροπολογίες ώστε να ενισχύσουν τον χαρακτήρα ανταγωνισμού των διατυπώσεων αυτών. Συμφωνεί με τις παραγράφους 7 και 8 που είναι πραγματικές διατάξεις περί ανταγωνισμού. Καταρχήν και τελειώνω, συμφωνούμε με την συνολική πρόθεση και κατεύθυνση της προτάσεως, ίσως για κάποιες λεπτομέρειες από πλευράς της και ηγετρίας να κατατεθούν κάποιες τροπολογίες, και ευχαριστεί και τον κύριο Κράμερ για την εξαιρετική συνεργασία. Μάισνερ. Α, θα συμφωνήσω κι εγώ. Ευχαριστώντας τον εισηγητή για το έργο του και για την συνεργασία μέχρι τώρα και εγώ εκπροσωπώ ε, τον σκιώδη εισηγητή που είναι σήμερα απόν φαίνεται να δημιουργείται μια τάση ολόκληρη ο κύριος ε, Τεξτέξ μου ζήτησε να σας ε, πω λίγα πράγματα γενικότερα, δεν ταυτίζονται με τις παραγράφους σας. Αφενός θεωρεί ότι είναι σημαντικό και θα υποβάλει τροπολογίες. Το κύριο θα πρέπει να είναι η προσπάθεια συνολικής δημιουργίας της ε, ενιαίας αγοράς και να μην δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ένα τρόπο μεταφοράς. Δεύτερον, θεωρεί ο σκιοδησηγητής ότι πρέπει να ερωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει μια επισκόπηση όλων των κρατικών ενισχύσεων που έχουν εγγυηθεί χώρες και μια επισκόπηση ενισχύσεων που δίνονται τώρα στις δημόσιες μεταφορές, και αυτό είναι ε, επιθυμία του κύριου Στέρξ. Για τα δικαιώματα των επιβατών, παρόλο που είναι σημαντικά, θεωρεί ότι δεν είναι απαραίτητο να μνημονευτούν εδώ, διότι δεν θεωρεί ότι εντάσσονται στην πολιτική ανταγωνισμού. Απλώς σου μεταφέρω την άποψη αυτή. Επίσης θεωρεί ότι πρέπει να περιληφθεί και αυτή η αναδιατύπωση του πακέτου των σιδηροδρόμων, αυτό το recast, που είναι σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την ε, ολοκλήρωση της πολιτικής ανταγωνισμού. Πέμπτο, από φέτος ισχύουν οι νέοι κανόνες για το καμποτάζ στις οδικές μεταφορές. Και δεν θα ήταν σωστό μήνυμα για το άνοιγμα της αγοράς, διότι έτσι με τις διατάξεις αυτές μειώνονται οι δυνατότητες της ε, εφαρμογής του καμποτάζ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενία Αγορά. Για τις ταχυδρομικές υπηρεσίες ο Στέρξ θεωρεί ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί η αγορά στον τομέα αυτό και θεωρεί σημαντικό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βελτιώσει την εποπτεία της για τις κρατικές ενισχύσεις. Το τελευταίο, τα είπε συχνά ο κ. Στέρξ επίσης, θεωρεί σημαντικό να υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για τα λιμάνια. Αυτά έχουν λεχθεί κάτι επανάληψη ότι χρειάζονται αυτές οι guidelines που δεν υπάρχουν ακόμα, δεν έχουν υποβληθεί ακόμα και αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό. Αυτά για την ώρα από τον κύριο Στέρξ. Ευχαριστώ κύριε Φώστερ. Θα είμαι και εγώ λακωνική. Δεν ξέρω πού είναι και ο δισηγητής νομίζω απουσιάζει. Πάντως ε, ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε ο κύριος Κράμερ. έχω κάποιες απορίες. Όλοι είμαστε υπέρ του θεμητού και δίκαιου ανταγωνισμού. Αλλά όταν εξετάζουμε χρηματοδότηση και χρέωση υποδομών και διάφορα άλλα θέματα και μιλούμε για τα είδη των μεταφορών, τα μέσα μεταφορών που χρηματοδοτούνται, που επιχορηγούνται, ορισμένα όντως επιδοτούνται συνεχώς, όπως οι σιδηρόδρομοι και κάποια άλλα μέσα μεταφοράς, για το σημείο 4 mm. είχαμε σοβαρές ανησυχίες και εμείς για τις καθυστερήσεις ε, στα αισθήματα αποζημίωσης και είδαμε με λεπτομέρειες κάποια δικαιώματα επιβατών στους σιδηροδρόμους. Δεν ξέρω, ίσως Καλύτερα να υπάρχει ένα ειδικό έγγραφο για τα δικαιώματα επιβατών σιδηρόδρομου και όχι τέτοιε λεπτομέρειε στη δική σας γνωμοδότηση. Στο σημείο 7 αναφέρθηκε το θέμα των ε, εταιριών low cost. Φυσικά θέλουμε μια υγιή πολιτική αεροπορία και μεγαλύτερη επιλογή των επιβατών ανάμεσα στις αεροπορικές εταιρείε ε, low cost και όχι τόσο φθηνών. Είναι θέμα επιλογή καταναλωτού. Τώρα, αν θα πρέπει να ισχύουν ειδικέ προποθέσει για ορισμένες επιχειρήσεις σε ορισμένα αεροδρόμια, το έχουμε ξανασκεφτεί και ξανασυζητήσει. Θα πρέπει να το φροντίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποφευχθεί αθέμετο ανταγωνισμό. Και έχω και μια επιφύλαξη για την παράγραφο 8, ίσω φταίει η μετάφραση. Καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμόζεται στον τομέα των αερομεταφορών η διευθέτηση που αφορά κρατική ενίσχυση σε ορισμένε περιπτώσει που βασίζεται στην αρχή first time, last time. Τι εννοείται, τα slot, τι χρονοθερίδε, τι θα πει first time, last time, last time και κρατική ενίσχυση. Νομίζω ότι υπάρχει απελευθέρωση πια στι αερομεταφορέ. Δεν ενισχύονται με επιχορογήσεις. Α, η Αιλιτάλια, που υπό ειδικέ προποθέσει για να συνεχιστεί η επιβίωση της, το ίδιο και με την Ολυμπιακή. Πάντως γενικώ έχουμε αυστηρούς κανόνες και απαγορεύονται κανονικά οι κρατικές ενισχύσεις στην αεροπορία. Αλλά ίσως ε, φταίει η αγγλική μετάφραση που δεν καταλαβαίνω την τροπολογία 8. Την ε, παράγραφο 8. Πάντως ε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξετάζουμε την γραμμοδότηση. Καλώς. Πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα κύριε Κράμερ να επανεξετάσετε το θέμα του αθέμητου ανταγωνισμού στις, στην αυσιπλοεία. Γιατί μία νταλίκα μπορεί κάλλιστα να περάσει τα σύνορα χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά τη συμπλήρωση των εντύπων στα τελωνία αν όμως προσπαθεί κανείς να μεταφέρει διαθαλάσσεις εμπορεύματα, εκεί εμπλέκεται σε ένα φοβερό χαρτομάνι και έχει τεράστια προβλήματα και με τις τελωνιακές διατυπώσεις. Από αυτή την άποψη των ε, συνθηκών ε, ισότιμου ανταγωνισμού θα πρέπει να το εξετάσουμε, γιατί οι θαλάσσιες μεταφορές επιβαρύνονται πολύ μεγαλύτερη γραφειοκρατία από ό,τι άλλα μέσα μεταφοράς. Και για το first, time, last time, όντως ε, κύριε Φώστερ, είναι υπενιγμός για ορισμένες ε, εταιρείε που τελευταία φορά κρατικής ενίσχυσης για αυτές δεν είναι και πολύ τελευταία. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά ξανά στον εισηγητή. Κυρία Μπρόντς, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζουμε βεβαίως την έκθεση που μας παρουσίασε ο εισηγητής και νομίζω ότι περιλαμβάνει και όλα τα κεντρικά στοιχεία της περσινής πρότασης. Ε, ο ανταγωνισμός στον τομέα των μεταφορών είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαρκώς προσπαθεί να εξυγχρονίσει το νομοθετικό ρυθμιστικό ε, πλαίσιο ε, και τους κανόνες ε, του ανταγωνισμού. Βεβαίως τα ζητήματα κρατικών επιχορηγήσεων οπωσδήποτε είναι πάντα στην πρώτη γραμμή για την περίοδο 2000-2009 και είχαμε σημαντικές εξελίξεις αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και στον ε, τομέα των κρυφών κρατικών επιδοτήσεων έχει γίνει πάρα πολλή δουλειά. Βεβαίως σημειώνουμε ε, όλες τις προτάσεις που γίνονται στην ε, έκθεση στα πρώτα τμήματα της ε, έκθεσης ε, θα μας ε, οδηγήσουν σε συνεργασία γιατί θέλουμε να τα ξανασυζητήσουμε και ε, επίση όσον αφορά τις εταιρείες low cost, χαμηλού κόστου και όσον αφορά τις κρατικές επιδοτήσεις ε, κρυφές ή φανερές, οπωσδήποτε ε, είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και το οποίο βεβαίως θα μας οδηγήσει σε κάποιες κυρώσεις. Μάικλ, να απαντήσεις. Φαίνεται πως δεν είμαστε σε θέση να επιβάλλουμε τον θέμητο ανταγωνισμό. Ορισμένοι ε, πληρώνουν φόρο καυσίμων, άλλοι όχι και ούτε καθεξής. Πρόκειται λοιπόν για αποδυνάμωση. Εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε διστακτικοί. Πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειες όλοι και τα τρία θεσμικά όργανα, ώστε να επιτευχθεί ο θεμητός ανταγωνισμός. Τώρα για ορισμένες ερωτήσεις, για το first time, last time, νομίζω ότι διευκρινίστηκε 27 φορές last time, καταλαβαίνεις τι ενός πρόκειται. Με τα έντυπα είχαμε νομίζω κάποτε μια έκθεση που έλεγε ότι έχουμε τα ίδια έντυπα για όλους τους τρόπους μεταφορών. Είπαμε να μην υπάρχει διαφορετικό έντυπο για τα τρένα, διαφορετικό για τα φορτικά, διαφορετικό για τα λιμάνια. Να υπάρχει ένα ενίο έντυπο και νομίζω το έχουμε αποφασίσει εδώ και μένει να υλοποιηθεί. για πολλά από αυτά που είπατε εκ μέρους του κυρίου Στέρξ είναι σωστά. Έχουμε σημαντικές επιτυχίες στον αυτοκινητόδρομο και στα αεροπλάνα γιατί είναι ανοιχτά τα σύνορα αλλά στο σιδηρόδρομο είναι όλα περιορισμένα. Γιατί? Γιατί στην ουσία είναι τα τελευταία καταφύγια του εθνικισμού. Εμείς όμως θέλουμε να περάσουν περισσότερα εμπορεύματα στο τρένο. Έχει λοιπόν πολλή δουλειά να γίνει ακόμα. Τελευταίο θέμα θα ήταν καλό να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το επίπεδο εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει επιτύχει το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο στη Γερμανία και όφωνα μάλιστα στις 18 ε, Δεκεμβρίου 2009. στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο που, όπου συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των 16 ε, ομόσπονδων χωρών ε, της Γερμανίας. Γι' αυτό και, εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ και χαίρομαι για τη συνένεση που ανακοινώσατε, κύριε Κούν. Σας ευχαριστώ, Μάικλ. Κλείσε το μικρόφωνο σου, Μίκαελ. Κλείσε το μικρόφωνο σου. Χρονοδιάγραμμα. 6 Οκτωβρίου λίγη η, τροπολο... η προθεσμία για τις τροπολογίες. 8 Νοεμβρίου θα εξετάσουμε τις τροπολογίες και θα ψηφίσουμε στις 9 Νοεμβρίου στην Επιτροπή Μεταφορών, ώστε να προλάβουμε την ε, ψηφοφορία στην ΕΚΟΝ στις 30 Νοεμβρίου. Η έκθεση έχει προβλεφθεί για την Ολομέλεια του Δεκεμβρίου, ενδεχομένως. Διορία για την κατάσταση τροπολογιών η 6η Οκτωβρίου. Αυτά και να περάσω στο τελευταίο σημείο τη ημερήσια διάταξη. Προηγουμένω όμω να πω σε όσου μεταβούν στην Αυστρία, Σλοβενία και Κροατία αύριο να τους ενημερώσω ότι θα γίνει απεργία, δυστυχώς, οπότε θα πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο για να πραγματοποιήσουμε την αποστολή. Ραντεβού στις 7 στο Κάρτο Μιντή να πάρουμε το τρένο για τη Φραγκφούρτη και από τη Φραγκφούρτη θα πετάξουμε στο Γκράτς. Θα ήθελα η γραμματεία να μου πει ποιοι θα συμμετέχουν στην αντιπροσωπεία. Πάντως, άλλο τρόπο δεν έχουμε να πάμε στη Φραγκφούρτη παρά μόνο σιδηροδρομικός. Αύριο στι Βρυξέλλε δεν θα κυκλοφορήσουν ούτε τα μέσα μαζική μεταφορά, οπότε και θα έχουμε πρόβλημα ακόμη και να μεταβούμε στη Γκάρντου Μιντή. 7 το πρωί πάντως ραντεβού στο Γκάρντου Μιντή για να πάρουμε το τρένο για τη Φραγκφούρτη 7 και 25. Περνάμε στην έκθεσή μου για τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία για τον τουρισμό. Θα σας παρουσιάσω το σχέδιο έκθεσης και θα κάνω κάποια σχόλια. Είμαι υπέρ της πρότασης του κανονισμού που προβλέπει ότι η διαδικασία λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να συνοδεύεται από στατιστικές που θα αντανακλούν τις ε, τάσεις στον τουρισμό κτλ. Επίσης θέλουμε συγκρίσιμα δεδομένα. Τα συγκρίσιμα δεδομένα είναι σημαντική βάση για την εφαρμογή της πολιτικής μας για τον τουρισμό. Έχω όμω δύο ανησυχίες ό,τι αφορά τον κανονισμό. Καταρχήν, η Κομισιόν θα μπορεί να τροποποιήσει σημαντικά σημεία του κειμένου, όπως τους ορισμούς, τα θέματα και τα χαρακτηριστικά των απαιτωμένων πληροφοριών, χρησιμοποιώντας αυτό το μέσο των ε, νομοθετικών πράξεων κατά εξουσιοδότηση. Και μια και πρόκειται για μη νομοθετική διαδικασία, προτείνω διάφορες τροπολογίες προκειμένου να περιοριστούν οι αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα και με την θέση του Κοινοβουλίου για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Επίσης, η πρόταση αυτή δεν προβλέπει τα TSAs, δορυφορικούς λογαριασμού για τον τουρισμό, που περιλαμβάνουν στατιστικές τουρισμού και κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες που δείχνουν τα αποτελέσματα του τουρισμού στις θέσεις εργασίας και την οικονομία. Οπότε προτείνω μια διάταξη προκειμένου τα κράτη-μέλη να μπορούν να καταρτίζουν πειραματικές μελέτες για τους δορυφορικούς λογαριασμού τουρισμού που θα εξετάζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εν ανάγκη θα υποβάλλεται νομοθετική πρόταση για υποχρεωτική εφαρμογή των δορυφορικών λογαριασμών για τον τουρισμό. Τέλο προτείνω πειραματικά προγράμματα προκειμένου να δημιουργηθεί ένα σύστημα για την σύμπτυξη δεδομένων και την ενοποίηση των δεδομένων που δίνουν τα αποτελέσματα του τουρισμού για το περιβάλλον. Φαίνεται ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφωνούν και σε ό,τι αφορά τον περιορισμό των κατεξουσιοδότηση πράξεων και την προοδευτική ε, εισαγωγή κατάρτιση δορυφορικών λογαριασμών για τον τουρισμό. Οπότε είναι σκόπιμο να διερευνήσουμε την πιθανότητα ε, πρόορης με το Συμβούλιο αν συνεχιστεί αυτή η σύμπνοια. Ζήτησαν το λόγο ο κύριος Φιντάντσα και η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν ε, να, συγχαρώ, να σας συγχαρώ, κύριε Πρόεδρε, για το σχέδιο αυτό της έκθεσης που ευθυγραμμίζεται και με τις δικές μας προσδοκίες. Θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμός ε, του 1995. θα πρέπει να εξυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί στις ε, εξελίξεις της αγοράς, αλλά και τις νέες τουριστικές συνήθειες. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στα βασικά σημεία του νέου αναθεωρημένου κανονισμού. Υπάρχει το θέμα της κατεξουσιοδότησης ε, πράξεων, το πιο επίμαχο ζήτημα. Και νομίζω ότι η θέση του Συμβουλίου είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Ζητήματα όπως ε, οι, προ... ορισμοί, τα θέματα, ε, τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν τα στατιστικά στοιχεία, όλα αυτά θα πρέπει να υπόκειται στην συνηθισμένη νομοθετική διαδικασία και να μην υπόκειται στη διαδικασία κατά εξουσιοδότηση πράξεων. Επίσης, ε, είναι σημαντική η μνήμα της εισαγωγής των δορυφορικών λογαριασμών, γιατί είναι ένα επιπλέον στοιχείο που βελτιώνει την κατάσταση και δίνει μια ευρύτερη εικόνα για τα συναφή με το τουρισμό θέματα, όπως ε, τις επιπτώσεις του τουρισμού στην οικονομία, στην απασχόληση και στο περιβάλλον. Οπότε είναι εύλογο που επιμένουμε στο θέμα αυτό των δορυφορικών λογαριασμών που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον αναθεωρημένο κανονισμό. Υπάρχει και ένα άλλο σημείο, το θέμα των ε, επισκέψεων που αναφέρεται στον κανονισμό. Εγώ θα ήθελα στο δεύτερο παράρτημα να περιληφθεί το τμήμα 3 για τις ημερήσεις αυτές επισκέψεις. Αν όμως αυτά τα μονοήμερα ταξίδια θα πρέπει να δούμε αν είναι όντως τουριστικά ή απλώς ε, εντάσσονται στην άσκηση της ελευθερίας διακίνησης. Να δούμε τι θα πει τέτοια μονοήμερη επίσκεψη. Για να δούμε τι εμπίπτει σε αυτόν τον ορισμό και τι όχι. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτό το σημείο και να δούμε τι πραγματικά σημαίνει αυτό το μονοήμερο ταξίδι, ή ημερήσιες επισκέψεις, για να μην επιδέχεται αυτή η έννοια στις ερμηνείας στις διάφορες χώρες. Προσπάθησα να συγκρίνω τα διάφορα τμήματα του κανονισμού και θεωρώ ότι είναι σκόπιμο στο 2-2 εκεί που γίνεται λόγος για τα, τις ατομικές δαπάνες του τουρίστα και όχι μόνο για τις μεταφορές, αλλά και για την διανυκτέρευση, παραμονή στο ξενοδοχείο κτλ. Να ληφθούν υπόψη και οι δαπάνες ε, της διατροφής. Δηλαδή, εάν έφεγε κανείς ε, σε εστιατόρια ή κάπου αλλού, γιατί και αυτό μπορεί να είναι καλός ε, δείκτης, σημαντικός. Πάντως, νομίζω ότι υπάρχουν περιθώρια καλά, έτσι ώστε σε πρώτη ανάγνωση να επιτύχουμε συμφωνία με το Συμβούλιο και νομίζω ότι άνετα μπορούμε να ε, προσανατολιστούμε προς αυτόν τον στόχο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μάισεν. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος του σκιώδου κ. Ούτσας, που θεωρεί πολύ σημαντικό το θέμα, ενδιαφέρεται για τον τουρισμό και θα προτιμούσε να γίνει συνάντηση των σκιωδών εισηγητών με τον εισηγητή πριν από την κατάθεση εκθέσεως. Ο κ. Ούτσας τονίζει ιδιαίτερα, διακόπτει ο πρόεδρος, ο εισηγητής που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής είναι, έχει αρκετά φορτωμένο πρόγραμμα και έχει γίνει εισηγητής μόνο και μόνο επειδή κανένας άλλος δεν ήθελε. Λοιπόν, αυτό τα λέω και μεταφέρετε τα στον κύριο Ούτζιας. Αγαπητέ πρόεδρε, το γνωρίζουμε καλά αυτό. Και γι' αυτό είπα ότι ο κύριος Ούτζιας το γνωρίζει και, αυτό, και αυτός. Αλλά είπα ότι ενδιαφέρεται πολύ για το θέμα και χαίρεται ιδιαίτερα για την συνεργασία η οποία θα συμβεί. Ε, τώρα για την πρώτη τροπολογία που θεωρεί σημαντική διότι δείχνει ποια είναι η σημασία του τουρισμού και ποια είναι η συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη και στην απασχόληση και ότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο, ιδίω για ορισμένε απομακρυσμένες περιοχές Ο κ. Σούτζας είναι και αυτό ε, νησιώτης, που λόγω των γεωγραφικών συνθήκων δεν έχουν άλλη δυνατότητα να προσφέρουν πολλή απασχόληση. Εκεί λοιπόν είναι σημαντικό να ε, συλλέγονται τα στατιστικά αυτά δεδομένα, ώστε να μπορούμε να δούμε πώς ε, κινείται η ανάπτυξη, τι ε, μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί και να βελτιωθεί επίσης η απασχόληση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προτάσεις της Κομισιόν, σε σχέση με τις εποχικές διακυμάνσεις. Είναι επίσης σημαντικό στην ανάλυση αυτή να δούμε πώς μπορούν να παραταθούν οι σεζόν. Η στατιστική ανάλυση θα παίξει σημαντικό ρόλο για να δείξει τι μπορεί να γίνει στις επιμέρους περιφέρειες ή περιοχές, ώστε περισσότερα από τα έσοδα του τουρισμού να διατεθούν μετά υπέρ των περιοχών αυτών. Επίσης ο κ. Σούτζας χαίρεται για την πρότασή σας κύριε Πρόεδρε και εισηγητά για τον, που, ταιριάζει και με τον μεγαλύτερο ρόλο που παίζει τώρα το Κοινοβούλιο ως συνομοθέτης και σε γενικές γραμμές ο κύριος Ούτζας σας επενεί και σας ενισχύει έχοντας έστω εκφράσει στην αρχή την επιθυμία για περισσότερη ακόμη συνεργασία μαζί σας. Μάλιστα, ευχαριστώ. Κομισιόν, κύριε Δε Μούντερ. Α, εσύ, Μίχαελ Κράμερ. Ναι, ακριβώς. Γιατί τα λέει όλα ο κύριος Κούν και χωρίς μικρόφωνο. Αυτές οι στατιστικές του τουρισμού είναι σωστό. Εκεί περιλαμβάνονται και όλες, όλοι οι τρόποι μεταφοράς, αλλά όχι το ποδήλατο, που ωστόσο έχει σημαντική αύξηση τζίρου 20% τον χρόνο εδώ και 20 χρόνια. Άλλωστε είναι σημαντικό, σημαντικό να ενισχυθεί ο τουρισμός με ποδήλατο, ο οποίος ποδηλάτης, ε, το λέω και το ξαναλέω, δαπανά και περισσότερα από τον αυτοκινητιστή, διότι έχοντας ποδηλατήσει μια ολόκληρη ημέρα και φτάνοντας στον προορισμό του κουρασμένος δεν θα σκεφτεί να ε, τσιγκουνευτεί τα ένα και τα δύο ευρώ για να φάει ή να πιει κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ βέβαια και για την εργασία που έκανε ο εισηγητής, έστω και αν ε, ανέλαβε την έκθεση αυτή επειδή κανείς άλλος δεν την ήθελε. Ευχαριστώ ο Μιχαήλ. Πράγματι, ορισμένες φορές είναι υποχρεωμένος κανείς να κινηθεί. Ο κύριος Ντεμούντερ. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί εργαστήκατε επ' αυτού του θέματος. Και βεβαίως να σας ευχαριστήσω και για την έκθεση που ετοιμάζετε. Θα γνωρίζετε φαντάζομαι ότι λίγο μετά την ε, θέση σε ισχύ της ε, συνθήκης της Λαβώνας ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το, θέμα αυτό και επομένως οι προτάσεις μας βασίζονται και στις εξελίξεις όσον αφορά τις περιφερειακές συμφωνίες όσον αφορά τις πράξεις κατεξουσιοδότηση μπορούμε να δεχτούμε διεθνείς τροπολογίες ε, κυρίως τροπολογίες 2, 3, 5 και 10 και επίσης 11 ε, έως 16. Υπάρχουν όμως και κάποιες εξαιρέσεις, ένα θέμα το οποίο αναφέρθηκε από τον κύριο Φιντάντσα, δηλαδή το θέμα των ειδικών ε, των ειδικών ε, επισκέψεων. Ε, νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να συμπεριληφθούν. Παρόλα αυτά όμως στον κανονισμό θα γίνει αναφορά τουλάχιστον ε, με αναφορά σε σχέση με τις στατιστικές τουρισμού. Ο λόγος για τον οποίο προτείναμε τον νέο κανονισμό ήταν ε, να βοηθήσουμε ε, τον τουρισμό παρουσιάζει μεγάλο βάρος ο τουρισμός στα έπα όλων των χωρών και επομένως είναι πολύ σημαντικός για να τον ε, αγνοήσουμε. Ε, όμως τα μηνύματα που έχουμε από τα κράτη-μέλη είναι ότι ακόμα σε αυτή τη φάση δεν είναι έτοιμα τα ε, κράτη-μέλη. Επομένως, καλωσορίζουμε και την τροπολογία ε, για προσθήκη ενός τμήματος 3 στο παράρτημα 2. Δεν ξέρω βέβαια αν το Συμβούλιο θα το δεχτώ, αλλά δεν μπορούμε εμείς να το καθαρίσουμε τη θέση του. Επίσης, θα μπορούσαμε εν είδη συμβαστικής λύσης να το συμπεριλάβουμε ε, στις στατιστικές τουρισμού αργότερα. Αργότερα ενδεχομένω ε, στην επόμενη φάση. Και έτσι να αναγνωριστεί και η δυνατότητα ε, η σημασία του θέματος αυτού. Τώρα, όσον αφορά τώρα την περιοδικότητα της συλλογή των δεδομένων, όσον αφορά το επίπεδο λεπτομέρειας και όσον αφορά ε, του, τις διορίες ε, μεταφοράς των δεδομένων, εκεί ε, τα κρατημέλη δεν είναι ακόμα έτοιμα και, μας θα κριθεί το ποιες παράμετροι θα μετρηθούν αυτού του είδους μας επισκέψεις δεν φαίνεται ε, να να θέλουν οι περισσότεροι ε, να τις βάλουμε στις στατιστικές τουρισμού, αλλά να ακολουθήσουμε ε, τις λοιπές στατιστικές. Εάν το Συμβούλιο συμφωνήσει βέβαια ότι αυτές οι επισκέψεις μπορούν να μπουν στις στατιστικές τουρισμού, τότε είναι διαφορετικά. Το, το σημαντικό είναι να βρούμε από κοινού ποια είναι τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συλλεχθούν. Ε, τροπολογίες, ε, ε, τροπολογία α7, συμφωνούμε ότι αφορά ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, αλλά θα θέλαμε μια διαφορετική διατύπωση παρόμοια με τη διατύπωση της τροπολογίας 5. Και στην τροπολογία 10 για τις ε, διορίες ε, μετάδοση δεδομένων εκεί που γίνεται λόγος ε, στην παρακολούθηση κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων και εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξουσιοδότηση. Σχετικά με τις κατεξουσιοδότηση πράκτης μπορούμε να δεχτούμε τις αρχές, να δεχτούμε τα θέματα επί των αρχών, να, επί της αρχής, συγγνώμη, να ε, και μπορούμε να δεχτούμε κάποιες τροπολογίες όπως είπα και προηγουμένως. Κατά τα λοιπά, ε, υπάρχουν και κάποια σημεία τα οποία ε, μπορούμε περαιτέρω να διερευνήσουμε, άρθρο 3, 4 και 7, τροπολογίες 5, 6, 10. Τώρα όσον αφορά την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και η Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων θέλουν ε, τέτοιου είδους στατιστικές, όχι μονάχα η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Επομένως, είναι θετικό που ο εισηγητής κάνει μια τέτοια αναφορά ε, και αναφέρεται και σε διασύνδεση με τις ε, υπόλοιπες μελέτες όσον αφορά τις τροπολογίες ε, για περιοδική αναφορά στο Κοινοβούλιο βεβαίως συμφωνούμε. Όσον αφορά το τμήμα το οποίο αναφέρεται στην, στις επιπτώσεις του τουρισμού στο περιβάλλον παραπέμπομαι στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 2007 που αναφερόταν σε αηφόρο ε, και ανταγωνιστικό τουρισμό. Άρα οι αρχές που αναφέρονται εκεί είναι αυτές με τις οποίες συμφωνούμε, αλλά μπορούμε να ε, συμφωνήσουμε ε, και με την άμεση διατύπωση στην παράγραφο 4 του νέου. Βεβαίω, κυρίω και όσον αφορά τι πράξεις ε, κατά εξουσιοδότηση, είναι γεγονός ότι περιμένουμε και τη θέση του Συμβουλίου και το λέτε κι εσείς. Όσον αφορά την, ε, ε, την ταχύτητα με την οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το σφάκελος αυτός, συμφωνούμε. Συμφωνούμε και ότι θα πρέπει έστω και ατύπως να καθίσουν, να συζητήσουν και τα τρία θεσμικά όργανα έτσι ώστε να αμπληθούν όσο γίνεται οι διαφορές. Αυτά ήθελα να σας πω και αυτές είναι οι παρατηρήσεις μου σχετικά με την έκθεση του κυρίου ε, Σίμψον. Όσον αφορά τα, σχόλια τα οποία ανέφεραν κάποια από τα μέλη της Επιτροπής, ήδη απήντησα σε ορισμένες από τις ερωτήσεις. Όσον αφορά τώρα τις ε, δαπάνες, ναι, βεβαίω στο σύνολο των δαπανών, στη συλλογική δαπάνη δηλαδή, συμπεριλαμβάνεται και η τροφή. Όσον αφορά τώρα από την σκοπιά της συλλογής ε, δεδομένων, ε, ή θα πρέπει να μειώσουμε τις ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν ή ε, θα πρέπει να βασιστούμε σε ένα πιο αξιόπιστο συνολικό αριθμητικό στοιχείο. Πάντως, όπως είπα και προηγουμένως, μπορούμε να δεχτούμε ενδεχομένω τις ε, τροπολογίες αυτές, περιμένοντας βέβαια να δούμε και τι θα κάνει και το Συμβούλιο. Όσον αφορά... Ε, την εποχικότητα ε, ε, βεβαίως ε, ε, έχουμε την εποχικότητα δεδομένη από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς τα στοιχεία για τις στατιστικές μας έρχονται από τα ξενοδοχεία και τα υπόλοιπα καταλήμματα και έρχονται αναμίνα. Στο παράρτημα 2 αναφέρουμε ε, τα ταξίδια των ε, κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τρόπο μετακίνησης και ανά ταξίδι ε, και επομένως στοιχεία υπάρχουν, απλώς δεν μπορούν να τα δώσουν όλα τα κράτη-μέλη γιατί δεν έχουν ακόμα το σωστό τρόπο τυποποίησης. Θα πρέπει να περιμένει λίγο η Eurostat. Όσον αφορά τους τρόπους, τα μέσα, τα μεταφορικά μέσα, η Επιτροπή γνωρίζει την αυξανόμενη σημασία των ε, ε, ποδηλάτων, οργανωμένες ε, ποδηλατικές ας πούμε διακοπές ξέρουμε ότι κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος και οπωσδήποτε κάποια στιγμή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα στοιχεία που αφορούν το ποδήλατο. Απλώς ε, απλώς πολύ συχνά γίνεται αναφορά στο κύριο μέσο μεταφοράς, εννοώντας το μέσο με το οποίο φτάσατε στον προορισμό σας έστω και αν μετά χρησιμοποιεί κάποιος το ποδήλατο, καταγράφεται ως κεντρικό κύριο μέσο μεταφοράς ο, ο τρόπος με τον οποίο έφτασε, ε, με κάποιο, έφτασε στο, κεντρικό, στο κύριο προορισμό, δηλαδή το λεωφορείο, το αυτοκίνητο, το τρένο κτλ. Παρατήρησε ο μικροφόνου. Ναι, βεβαίως όταν ζητούμε ε, όταν ζητούμε στοιχεία για διατροπικότητα ε, ε, είναι λίγο πιο δύσκολο να καταγράψουμε τα στοιχεία. Όσον αφορά τώρα τις συνδυασμένες στατιστικές και την επίδραση που μπορεί να έχει ο, ο ένας τρόπος σε, κάποια άλλη, σε κάποιο άλλο στατιστικό στοιχείο. Είπατε ότι αυτοί που κάνουν ποδηλατικές εκδρομές ενδεχομένως μετά θα φάνε περισσότερο. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποτυπωθεί. Τώρα, εάν ε, και η αποστολή των στατιστικών στοιχείων και το Κοινοβούλιο συμφωνήσει ότι κάποια συγκεκριμένα στοιχεία θα πρέπει ε, να μεταδοθούν και να συμφωνήσει και οι, γενικοί, οι άλλες γενικές διευθύνσεις επιχειρήσεων και βιομηχανίας, τότε εντάξει, θα συμφωνήσουμε και εμείς. Τώρα για τα μονοήμερα ταξίδια. Ξόδησα πολύ χαρτί και χρόνο για αυτό το θέμα. και επίση τι να περιλαμβάνεται σε αυτό το θέμα της διατροφής λοιπά. Περιμένω πάντως τις τροπολογίες σας και τότε θα συνεννοηθώ με τους σκιώδες ηγητές και θα συζητήσουμε με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. 4 Οκτωβρίου λίγη διορία για τις τροπολογίες. Θα ψηφίσουμε στις 27 Οκτωβρίου στην Επιτροπή μας και κατά πάσα πιθανότητα στην Ολομέλεια τον Νοέμβριο. Οπότε στείλτε μέχρι τις 4 Οκτωβρίου τις τροπολογίες σας, να τις εξετάσω με τους σκιώδες ηγητές για να καταλήξουμε σε κοινή θέση, ώστε να αρχίσουμε μετά τις συζητήσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Και αν το Συμβούλιο και, το Κοινοβούλιο, αν το Συμβούλιο και η Επιτροπή συμφωνήσουν με το Κοινοβούλιο, είμαι σίγουρος ότι τα πράγματα θα πάνε να Πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και τον κύριο Τεμούλτερ. Διάφορα υπάρχουν. Όχι. Επαναλαμβάνω αυτό που είπα νωρίτερα. Ενημερώστε τα μέλη της αντιπροσωπείας που θα μεταβεί ε, στις ε, τρεις χώρες για την αλλαγή λόγω της απεργίας. Να μην πάρουν στο αεροδρόμιο να έχουμε ραντεβού 7 η ώρα το πρωί στην Καρτιμιντή. Η επόμενη μας συνεδρία θα γίνει στις 26 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη. Τρίτη 26 Οκτωβρίου στις 3 το απόγευμα στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ και τους Καλό σας απόγευμα.